Good morning. Καλή σα μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή Αναφορών σήμερα το πρωί και θέλω να καλωσορίσω ιδιαίτερα τους προσκεκλημένους μας. Σήμερα έχουμε δημόσια ακρόαση για την διαφάνεια και την ελευθερία πληροφόρηση ε, στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να σας δώσω πρώτα κάποιες πρακτικές πληροφορίες. Καταρχάς να απευθυνθώ στη στο Τμήμα Πολιτικής και να τους ευχαριστήσω για όλη τη δουλειά που έχουν κάνει. Επίσης, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση των εστονικών, φιλανδικών, λιθουανικών, πορτογαλικών, σλοβενικών και σλοβακικών. Και σας παρακαλώ να γνωρίζετε ότι η σημερινή ακρόαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο και θα ε, μαγνητοσκοπηθούν όλες οι παρεμβάσει. Και σήμερα λοιπόν έχουμε το θέμα διαφάνεια και ελευθερία πληροφόρησης, ε, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους πολίτες, διότι είναι θέμα απαραίτητο για να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία. Ε, εμείς που λαμβάνουμε αποφάσεις γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η σωστή ενημέρωση των πολιτών σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο σύστημα η θέση ισχύ του κανονισμού για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα έχει επιτρέψει στους Ευρωπαίους πολίτες να ζητούν πρόσβαση σε έγγραφα των ε, θεσμικών οργάνων και η συνθήκη της Λισαβόνα έχει υπογραμμίσει τη σημασία της ε, ανοιχτής ε, και διάφανης λήψης αποφάσεων καθώ και τη συμμετοχή των πολιτών. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει αυξανόμενο ρυθμό ετοιμάτων από πολίτες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θέλουν τώρα να είναι πιο καλά ενημερωμένοι σχετικά με τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και την ομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναπτύξει πολύ ενδιαφέρουσα νομολογία πάνω στο θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια. Η Επιτροπή μας επίσης έχει λάβει διάφορες αναφορές ε, στις οποίες οι πολίτες ζητούν, μάλλον αναφέρουν ε, έλλειψη διαφάνειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικά θέματα. Ωστόσο, υπάρχουν Κάποιε διαπραγματεύσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση, όπου τα θεσμικά όργανα και οι εθνικές αρχές ε, ισχυρίζονται ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο, στην θεμελιώδη ελευθερία των πολιτών ε, και την ανάγκη για πιστευτικότητα. Σήμερα λοιπόν ε, έχουμε αυτή την ακρόαση για την διαφάνεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο. Εύχομαι σε όλους μας επικοδομητική συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε δύο ομιλητές. Ε, την ε, καθηγήτρια Κέρτιν από το Πανεπιστήμιο της Φλωριντίας και ε, του Άμστερνταμ και τον ε, καθηγητή Σάνμπεργκ από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη. Θα μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους ε, εκ μέρους ε, του Τμήματος Πολιτικής ΓΑΜΑ. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά μαζί με τον συνάδελφό σας. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, θα μπορούσα να ξεκινήσω και ξεκινώ ευχαριστώντας για την ευκαιρία αυτή και την πρόσκληση να συνεισφέρουμε για αυτές τις παρουσιάσεις με αναλύσεις. Εστιαζόμαστε σε ένα θέμα όπου εργαζόμαστε επί αρκετά χρόνια ήδη και είναι πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα επικεντρωνόταν ιδιαίτερα στην δημοκρατία, στην διαφάνεια και στην βελτίωση της προσπελασιμότητας της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα, στα έντυπα. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να ανασκοπήσουμε και να δούμε τι, συνέβη, τι συνέβαινε από το 2009. Και προετοιμάζοντας μια τέτοια περιεκτική έκθεση είναι κάπως μια πρόκληση και σε σχέση και με την ομολογία που απέρευσε από το 10, από το 2009 θα αναφερθούμε σε κάποια από τα κυριότερα θέματα που εξέτασε το 10 ε, σε σχέση και με τις ρυθμίσεις ε, και ποιε απαιτήσει θα ίσως θα χρειαζόντουσαν επικαιροποίηση μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο αν δεν είναι πλήρως, πλήρες και αποτελεσματικό πως θα έπρεπε και θα έπρεπε να ανανεωθεί, να επικαιροποιηθεί. Θα μιλήσει για τις ε, προκλήσεις, ε, θα γίνει λόγος για τις προκλήσεις και τα θέματα που το Κοινοβούλιο πρέπει να προχωρήσει παραπέρα από πλευρά συστάσεων για το τι μπορεί να απορρέει από τις αναλύσεις που κάναμε και συντάξαμε. Και το πρώτο σημείο που θα θέλαμε να αναφέρουμε αφορά τον κανονισμό 1049 φυσικά και το γεγονός ότι με βάση τις αναλύσεις μας θεωρούμε ότι είναι ανεδαφικός ξεπερασμένος ο κανονισμός. Ολόκληρες δεκαετίες είναι παλαιός αυτός ο κανονισμός και σε σχέση και με τα θέματα τα οποία τίθενται δεν έχει επικαιροποιηθεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας και γνωρίζουμε όλοι επειδή οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το χαρτοφυλάκιο τροχοπεδήθηκαν επί πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 είναι και αυτή ξεπερασμένη και ανεδαφική. Τώρα σε σχέση με την ομολογία του 10 και γιατί θεωρούμε ότι έχει εκδώσει θετικές αποφάσεις το δικαστήριο σε σχέση με νομοθετικά θέματα. Υπάρχουν κύρια θέματα όμως στον κανονισμό που δεν καλύπτονται από την ομολογία και που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή του κανονισμού με τον ορθότερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ένα από τα θέματα αφορά την έννοια, την προσέγγιση του δημοσίου κοινού συμφέροντος. Ρόλο κλειδί έχει σε σχέση με τις σκέψεις πότε θα μπορούσε να εγκριθεί, η πρόσβαση σε τέτοια α, χαρτοφυλάκια και έγγραφα. Θεωρούμε ότι στην ομολογία του δικαστηρίου το θέμα του κοινού δημοσίου συμφέροντος ε, έμεινε πάρα πολύ λόγο και ήταν δύσκολο να πιστεί το δικαστήριο σε σχέση με θέματα όπως το περιβάλλον δημόσια υγείας, ε, δημόσιων κονδυλίων και λοιπόν θεωρούμε ότι το θέμα του δημοσίου συμφέροντος είναι κάτι που πρέπει να ρυθμιστεί και να επαναπροσδιοριστεί σε σχέση με τα θέματα νομολογίας. Ένα άλλο θέμα αφορά τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις, διότι ο κανονισμός βασίζεται σε δύο είδη εξαιρέσεων και οι υποχρεωτικές επιτακτικές εξαιρέσεις που απαιτούν από τα θεσμικά όργανα πάντα να αρνούνται πρόσβαση σε περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει επιζήμια επίπτωση σε συμφέρον, σε δημόσιο συμφέρον. Εδώ θεωρούμε ότι η εξέταση του δημόσιου συμφέροντος ως επιχειρήματος καμιά φορά πρέπει να είναι αναγκαία και σε σχέση με διεθνείς σχέσεις ε, από πλευράς ε, καθηγητού Κέρτη θα ε, υπάρξει αντίστοιχη τοποθέτηση επίσης. Και σε σχέση με την ομολογία πάλι σε σχέση με πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ή σε προσωπικό χαρτοφυλάκιο ενός ατόμου. Το άτομο να έχει δικαίωμα δηλαδή σε σχέση με πληροφορίες που το αφορούν το ίδιο όσον αφορά φακέλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο προστατεύεται συγκεκριμένα από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και όσον αφορά τη χρηστή διαχείριση. Βλέπουμε ότι από την ομολογία σε σχέση με το 1049 ως κανονισμό υπάρχουν περιπτώσεις νομολογίας που δεν ε, συμπεριλαμβάνουν τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα και άτομα αναζητούν προσωπικά την, τα δικά τους στοιχεία σε σχέση με φακέλους τους. Η πρόσβαση σε σχέση με τους φακέλους αυτούς δεν είναι κάτι που λειτουργεί όπως θα έπρεπε και αυτό θα έπρεπε ξεχωριστά να ρυθμιστεί από τα θεσμικά όργανα. Προτιμητέο θα ήταν σε σχέση με το πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης και σε σχέση με τις διοικητικές διατάξεις ρυθμίσεις που ελπίζουμε, ευελπιστούμε ότι μπορούν να, σε σχέση τώρα με το ξεπερασμένο πλαίσιο του, της ρύθμισης όσον αφορά και το θεσμικό πλαίσιο, διότι αυτή τη στιγμή μόνο προς το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή υπάρχει θέμα αναφοράς. Με βάση τη συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν ειδικό καθεστώς και μόνο σε σχέση με τις διοικητικές τους ε, υποχρεώσεις ε, και αρμοδιότητες ε, θα υπήρχε ένα περιθώριο. Αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι θεμητό και δεν δικαιολογείται. Αν δούμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το τι συμβαίνει, σε σχέση με μια τέτοια συνολική εξαίρεση θεωρούμε ότι δεν θα ήταν το πιο εύθετο. Δεν έχει αυτό καμιά σχέση με την νομισματική πολιτική. Και αυτά τα οποία βλέπουμε σε σχέση με τις ε, περιπτώσεις νομολογίας ότι το δικαστήριο είναι σχεδόν ελεύθερο από την υποχρέωση ε, δημόσιας προσπελασιμότητας και πρόσβασης από πλευράς των πολιτών σε σχέση για παράδειγμα με τον ανοιχτό χαρακτήρα δικαστικών διαδικασιών είναι μια αρχή που προστατεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας σε δύο αυτή τη στιγμή πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, αναλυφθεί από το Συμβούλιο σε αυτή τη φάση όσον αφορά τη Eurojust και το ESO όπου προτείνει το Συμβούλιο συνολικές τέτοιες εξαιρέσεις για τη Eurojust και το μελλοντικό, τη μελλοντική υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θεωρούμε ότι αυτό παραβιάζει τη συνθήκη είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε κάθετα να απορριφθεί, να το απορρίψουμε ως αίτημα. Τώρα, όσον αφορά <clears throat> τα έντυπα και έγγραφα, γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική νομοθεσία όσον αφορά το δικαστήριο σε σχέση με τη νομική γνώμη ή νομικές γνωμοδοτήσεις και ε, όσον αφορά τα κράτη-μέλη, πολύ καλές ε, περιπτώσεις αποφάσεων. Όμως ε, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες στο Συμβούλιο να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και οι κανονισμοί οι όσον αφορά τις κανονιστικές διατάξεις δεν έχουν επικαιροποιηθεί και γνωρίζουμε ότι όταν αφορά τέτοιου είδους ε, ε, νομικές νομοδοτήσεις ε, δεν συντάσσονται σε μια ανοιχτή δημόσια βάση και αυτό θα έπρεπε να επανεξεταστεί σε σχέση με έγγραφα των τριμερών διαλόγων αλλά επίσης και όσον αφορά τις αξιολογήσεις που συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώιμη φάση της νομοθεσίας και όπου έχει πρόσφατα δηλωθεί ότι θα μπορούσε εδώ να λειτουργήσει λειτουργήσει κάτι όσον αφορά την ένταξή τους μέσα στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να αποκατασταθεί διότι είναι μια σημαντική φάση νομοθετικών διαδικασιών όταν προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νομοθετική πρόταση. Η νέα διοργανική συμφωνία όσον αφορά καλύτερη νομοθετική ρύθμιση είναι μια καλή ευκαιρία για τους τριμερείς διαλόγους σε σχέση με το συναφές αυτό θέμα και φυσικά το θέμα των τριμερών διαλόγων αφορά και σε εκκρεμότητα υποθέσεις ή αποφάσεις. Ε, είναι σημαντική αυτή η πτυχή θεωρώντας ότι η πρακτική από πλευράς του Συμβουλίου, οι τοποθετήσεις ε, του Συμβουλίου και οι γνωμοδοτήσεις δεν δημοσιοποιούνται ως κανόνας ε, στο κοινό και δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτές ε, τις αποφάσεις. Θα πρέπει να δούμε σε σχέση με τη διαφάνεια τι μπορεί να απορρεύσει ώστε να μην απομείνει εκτός του πλαίσιου διαφάνειας αυτό το πεδίο. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας επ' αυτού που θα μπορούσε σε σχέση με το έγγραφο του Κοινοβουλίου να τύχει συνέχεια σε, από πλευρά τη επιτροπή η πρόταση που διατυπώνεται. Γιατί βρίσκονται θέματα εκτός του 1049. Πολλά έγγραφα δεν γίνονται απόλυτα ε, σωστά κατανοητά και δεν ερμηνεύονται με τον τρόπο που θα έπρεπε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να έχει υποδειγματικό ρόλο δίνοντας το καλό παράδειγμα και σε σχέση και με τα διοικητικά έγγραφα και αυτό είναι θέμα ιδιαίτερης επικαιρότητα και συσχετίζεται με το θέμα των γενικών ε, όρων και προϋποθέσεων. Και αυτό είναι κάτι που το δικαστήριο δημιούργησε υιοθετώντα αυτή την προσέγγιση που θεωρούμε ότι δεν έχει όμως κάποια βάση στον ίδιο τον κανονισμό. Τι σημαίνει αυτό στην πρακτική εφαρμογή. Στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε τεράστιους τομείς που είναι ελεύθεροι όσον αφορά την, ε, προσπελα, την ε, πρόσβαση με βάση την Γενική Αρχή Όρων και Προϋποθέσεων. Έτσι μπορεί κάποιος να βασιστεί στην προϋπόθεση ότι τίποτα δεν θα δημοσιοποιηθεί από όλα αυτά. Και αυτό ε, μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας και εργασιών. Και υπάρχει ίσως η δυνατότητα ότι τα διοικητικά θέματα αν συνεχίζονται έτσι υπό τον όρο ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις για τον τρόπο εργασίας και ιδιαίτερα όσον αφορά τις γενικές προϋποθέσεις και όρους που τώρα επεκτείνονται όσον αφορά το, τις δυνατότητες ED pilot και των παραβιάσεων που δεν είναι χαρακτηριστικά διοικητικά μεν θέματα αλλά εμπλέκουν και τα κράτη-μέλη επίσης και ιδιαίτερα αυτοί οι φάκελοι αφορούν ε, ε, λογισμικό υλικό που ήταν δημόσιο κατά το παρελθόν στα κράτη-μέλη και καθώς κατέληξε στα, στους φακέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εξαπίνης ευνηδίως άρχισε να εποφελείται από το ειδικό καθεστώς και έτσι αποκλείονται πλέον. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε σχέση με το ε, ότι συνέβαινε κατά το παρελθόν. Και τώρα στρέφαμε στην καθηγήτρια Κέρτιν, παρακαλώ. Thank you, um, Ευχαριστώ πολύ, Παϊβή. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία στα όσα ήδη υπόθηκαν και να υπογραμμίσω κάποια από τα συμπεράσματα της έκθεσής μας. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα της προστασίας δεδομένων, αλλά και στο θέμα των διεθνών σχέσεων, που είναι και τα δύο θέματα όπου υπάρχει παρέκκληση όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα. Υπάρχει σημαντική νομολογία και στα δύο αυτά θέματα. Αλλά ιδιαίτερα μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και μετά από την πρόταση της Κομισιόν να τροποποιήσει τον κανονισμό το 2008, είδαμε σημαντικές εξελίξεις στην πράξη, οι οποίες τονίζουν ένα από τα βασικά μας μηνύματα ότι ο κανονισμός είναι ξεπερασμένος. Όχι μόνο ως δίκαιο, αλλά και ως πρακτική. Όσον αφορά την προστασία δεδομένων, υπάρχει αρκετά παλαιά νομολογία και ιδιαίτερα η υπόθεση Λάγερ της Βαβαρίας, όπου έχουμε άρνηση πρόσβασης ε, στις ε, πληροφορίες ε, λόγω της προστασίας δεδομένων δημοσίων αξιωματούχων. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα αυτό υπό το φως των εξελίξεων έκτοτε. Αλλά αυτό αποτελεί παράδειγμα του πώς το δικαστήριο εξετάζει με μονομένα τις υποθέσεις, ενώ θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για πιο συνολική προσέγγιση, ώστε από τη μία να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά με προστασία των δεδομένων από την άλλη. Θα πρέπει όμως να εισαχθεί η έννοια του δημοσίου συμφέροντος ε, στην ισορροπία αυτή πρόβλημα υπάρχει, ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τα δεδομένα αξιωματούχων σε δημόσιο ρόλο. Το θέμα λοιπόν είναι ποιος εξετάζει τις ισορροπίες αυτές. Το δικαστήριο εξετάζει κατά περίπτωση ή μήπως υπάρχει ανάγκη για μια πιο συνολική προσέγγιση. με δημοκρατική ευθύνη του νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει αλλάξει η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Θα έχουμε ένα νέο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί η ισορροπία στο θέμα αυτό. Από ό,τι γνωρίζω κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα τομέα όπου θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Um, Δημόσια σχέσεις. Ο άλλο τομέα όπου πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί η ιδιαίτερη σημασία είναι η πρόσβαση σε πληροφορίε ε, στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Έχουν γίνει σημαντικές ε, τροποποιήσεις ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας από το 2009 και μετά και σε άλλη νομοθεσία. Ωστόσο η νομολογία δεν έχει αλλάξει. Το δικαστήριο περιορίζεται από τη διατύπωση του ίδιου του κανονισμού και από το γεγονός ότι οι διεθνείς σχέσεις είναι υποχρεωτική εξαίρεση στον κανόνα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της διαπραγμάτευσης διεθνών συμφωνιών και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Έχει αλλάξει η οπτική μας ε, λοιπόν όσον αφορά τις, δημόσιες, ε, τις διεθνείς σχέσεις και γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρξουν αλλαγές στον τομέα αυτών. Υπήρξαν υποθέσεις ε, στο δικαστήριο όπου έχουν προσφύγει μέλη ε, του Ευρωκοινοβουλίου κιόλα, ε, που δεν ε, είχαν τη δυνατότητα ως ευρωβουλευτές να έχουν πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες και έπρεπε να βασίζονται στις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στο κοινό. Αυτή βέβαια δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση. Θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα αυτό συνολικά στο πλαίσιο αναθεώρησης του κανονισμού. Και βέβαια, Δεν αρνούμαστε ότι δημόσιο συμφέρον είναι η πρόσβαση στα έγγραφα. Υπάρχει όμως σε κάποιες περιορισμένες περιπτώσεις ε, η πιθανότητα το δημόσιο συμφέρον να είναι η εμπιστευτικότητα. Δεν θέλουμε λοιπόν πλήρη διαφάνεια με αυτή την έννοια. Φτάνουμε έτσι στα συμπεράσματά μας, αλλά και στα βασικά στοιχεία της έκθεσής μας. Ποιες είναι οι προκλήσεις ε, που υπάρχουν και ποιες είναι οι συστάσεις μας για το μέλλον. Όπως ήδη είπε η Πάεβη, υπάρχει στασιμότητα όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά αυτό είναι λογικό καθότι έχει αλλάξει η νομική βάση με τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά έχει αλλάξει και η πρακτική των θεσμικών οργάνων. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να αναθεωρηθεί ο κανονισμός για την πρόσβαση στα έγγραφα. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αφήνουμε όλη την ευθύνη στο δικαστήριο. Και έτσι όλα θα εξαρτηθούν από τις προσφυγές στο δικαστήριο, αλλά και από την ε, αντίδραση των θεσμικών οργάνων. Το δικαστήριο δεν μπορεί να αναδομήσει το σύστημα Μπορεί να υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται, αλλά ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι ακόμα και όταν υπάρχει σαφής απόφαση από το δικαστήριο, και αναφέρω την υπόθεση Τούρκο, Υπάρχει αντίδραση από πλευρά των θεσμικών οργάνων, δεν θεσπίζουν τις απαραίτητε αλλαγέ και βλέπουμε ουσιαστικά επανάληψη της ίδιας υπόθεση στο δικαστήριο. Και ποιο ξέρει πότε θα έχει λίγο διαφορετική σύνθεση στο δικαστήριο και τελικά κερδίσουν τα θεσμικά όργανα. Ε, θεωρούμε λοιπόν, και το γράφουμε αυτό στην εκθεσή μας, ότι υπάρχει δημοκρατική ευθύνη από πλευράς του νομοθέτη. Δεν μπορεί ποτέ το δικαστήριο να υποκαταστήσει αυτή την ευθύνη. Και ο ε, Ευρωπαίος ε, Διαμεσολαβητής ε, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο θέμα αυτό. Δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν ένα σαφές νομικό πλαίσιο το οποίο να είναι σωστά προσαρμοσμένο στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ε, είναι ένα από τα βασικά μηνύματα που θέλουμε να σας μεταφέρουμε. Επίσης κάτι που δεν λέγεται αρκετά συχνά είναι ότι ο κανονισμός αυτός αφορά κυρίως ε, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά προέκταση ε, άλλους οργανισμούς, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Δικαστήριο ε, έχουν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογή. Κάτι τέτοιο μπορεί να αλλάξει μόνο με τροποποίηση της συνθήκης. Δεδομένου όμως του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δικαστηρίου, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό. Φυσικά υπάρχει ανάγκη για εμπιστευτικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Θα πρέπει όμως να επανεξεταστεί αυτό υπό το φως των εξελίξεων όσον αφορά τα καθήκοντά τους. αλλά και η ανάγκη αυτή μπορεί να προστατευτεί με κάποιες εξαιρέσεις όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφά τους. Θα μπορούσαμε, εάν υπάρχει το σχετικό ενδιαφέρον, να αναπτύξουμε το θέμα αυτό. Θα κλείσω όμως εδώ προς το παρόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας για αυτή την πραγματικά σαγηνευτική δουλειά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να είναι κανείς σε αυτήν την κοινοβουλευτική ε, επιτροπή όπου σε συνεργασία και με τη διαμεσολαβήτρια που ήταν εδώ χθε και ανταλλάξαμε απόψεις για κάποια από αυτά τα θέματα είναι λογική και συνεπής αυτή η απάντηση σε αυτό το συμβάν και από εσά. Το να είναι κανείς ε, Σουηδός είναι και κάποια εξαίρεση καμιά φορά. Ε, φέτος στην Σουηδία εορτάζουμε 250 έτη διαφάνειας και ανοιχτού χαρακτήρα από το νομοθέτημα της ελευθερίας του τύπου που έγινε πραγματικότητα το 1766 και θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη αυτό από πλευρά ε, Φινλανδού πολιτικού, η Φινλανδία και η Σουηδία ήταν μια χώρα τότε, τότε ήταν ιερέας και πολιτικός, καμιά φορά πολύ ενδιαφέρον αυτός ο συνδυασμός και εκείνος κατέσε εφικτό αυτός ο άνθρωπος στη Σουηδία να επιτύχει η έγκριση της ε, νομοθεσίας ελευθερίας του τύπου. 1766 οι σκανδιναβικές χώρες είναι καμιά φορά μια εξαίρεση και ευελπιστούμε ότι μπορούμε να εμπνεύσουμε όντας μια εξαίρεση και άλλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό τον ανοιχτό χαρακτήρα σας και το ανοιχτό πνεύμα σας και για το ότι είσαστε αυστηροί και τα είπατε ε, με τρόπο άμεσο. Τώρα στη συνέχεια Γιώνας Έμπεσον επικεφαλής ε, όσον αφορά τη σύμβαση Όρχος και επικεφαλής ε, του κέντρου της Στοκόλμης για το περιβαλλοντικό δίκαιο. Θα μας παρουσιάσει ακριβώς το έγγραφο αυτό, διότι προέρχεται από το Policy Department C και το θέμα είναι πρόσβαση στις πληροφορίες, συμμετοχή στις λήψεις αποφάσεις και πρόσβαση σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα στις διαδικασίες. Κύριε Έμπεσον, αγαπητέ Ιώνα, έχετε τον λόγο τώρα για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές που με προσκάλεσαν να μιλήσω εδώ. Βλέπετε τον τίτλο θα θέσω το θέμα αυτό της παρουσίασής μου ε, στο κέντρο ε, ενός περιβαλλοντικού πλαισίου και θα το συνδέσω με τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και την πρόσβαση ε, στην δικαιοσύνη. Αυτά τα θέματα είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους. Ένας λόγος που το θέτω έτσι είναι γιατί η πρόσβαση στην ε, ενημέρωση και στην πληροφορία ε, αναπτύχθηκε πολύ νωρίς, ε, πολύ πριν από άλλες ε, εξελίξεις. Η Σύμβαση του Άρχους είναι μια διεθνή συνθήκη όπου όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενα μέρη. Είναι μια μοναδική διεθνή συνθήκη όπου το ανθρωπιστικό δίκαιο και το περιβαλλοντικό δίκαιο συνδέονται στο πλαίσιό της. Και αυτό το μείγμα δεν ε, αντικατοπτρίζεται μόνο στο περιεχόμενο της σύμβασης, αλλά και στο μηχανισμό αναθεώρησης. Δημιουργεί δηλαδή ε, μια επιτροπή ε, διεθνούς συμμόρφωσης που στην οποία μπορούν να προσφύγουν και μέλη του κοινού, αλλά και κράτη-μέλη. Και αν δεν είχαμε αυτό τον μηχανισμό θα είχαμε πολύ λίγα να κάνουμε, θα επανέλθω σε αυτό. Σχεδόν 150 ε, ιδιωτικοί πολίτε, α πούμε, και ιδιωτικοί φορεί προσέφηκαν, αλλά μόνο δύο κράτη-μέλη. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή ε, ήταν ε, μια δημιουργία τη δεκαετία του 90, μια διεθνή ας πούμε εξέλιξη που οδήγησε στην ε, διακήρυξη του Ρίο από τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την ε, ανάπτυξη και το περιβάλλον. Όταν υιοθετούνται αυτέ οι διακηρύξει, ποτέ δεν ξέρει αν θα επιβιώσουν δύο εβδομάδε ή δύο δεκαετίε. Να, εδώ έχουμε μια διάταξη όπου πολλά χρόνια μετά είναι πολύ πολύ ζωντανή. Το βασικό στοιχείο τη δήλωση αυτή του Ρίο ε, συνδέεται με στοιχεία που αργότερα θα αντικατοπτριστούν και στο, στη ε, αλλά και στην, ε, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσβαση στην δικαιοσύνη και πρόσβαση στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση. Ε, τότε, στι αρχέ τη δεκαετία του 1990, υπήρξε και άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που οδήγησε σε αυτέ τι εξελίξει, που, που ήταν οι πολιτικέ αλλαγέ στην Ευρώπη. Όπου ε, ε, έννοιε όπω η κοινωνία των πολιτών, εκδημοκρατισμό, ε, περιβαλλοντικά ανθρώπινα δικαιώματα ε, μπήκαν στην ε, διεθνή αρένα και συζητήθηκαν, ε, έγιναν τμήμα του διεθνούς δικαίου και τμήμα των αποφάσεων με πρωτοφανή τρόπο πριν επισέλθω στην ίδια τη σύμβαση και στα δικαιώματα που παρέχει και που συνδέει την πρόσβαση στην πληροφορία με την συμμετοχή του κοινού, θα ήθελα να εξηγήσω κάποια από τη λογική για αυτέ τι εξελίξει. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε και στι διεθνεί εξελίξει και στι ευρωπαϊκέ εξελίξει ότι υπάρχουν κάποια επιχειρήματα υπέρ αυτών των πραγμάτων. Θα βρείτε κάποια από αυτά στο προήμιο τη σύμβαση του Άρχου και στην ε, ε, Ενωσιακή Νομοθεσία. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι η συμμετοχή του κοινού και η πρόσβαση στην πληροφόρηση βελτιώνει την προστασία την, ε, της υγείας και του περιβάλλοντος. Ε, λαμβάνονται καλύτερες ποιότητα αποφάσεις, ε, προωθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και αναπτύσσει και βασίζεται στην έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εφαρμόζει σε νέα πεδία και νέα πλαίσια, κάτι πολύ σημαντικό ενισχύει την νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καθώς και την δικαιοσύνη ε, την, που εμπεριέχουν. Προωθεί και είναι πολύ σημαντικό ε, την εμπιστοσύνη στις δημόσιες αρχές και την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που συνέντευγαν με το περιβάλλον. Το να δίνουμε το δικαίωμα ε, στο κοινό να συμμετέχει δεν σημαίνει ότι απεμπολούνται αρχές, ε, απεμπολούνται δικαιώματα των αρχών, αντίθετα νομοποιούνται αυτές οι αποφάσεις των αρχών ε, αυτή τη διαδικασία. Και συνολικά οδηγεί σε μια περιβαλλοντική ε, δημοκρατία. Η σύμβαση του Άρχους έχει σαν στόχο, επίσης, να σας το υπενθυμίσω, παρότι δεν συντάχθηκε ως Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέλει να δημιουργήσει και δικαιώματα για τους πολίτες, και το ξεκαθαρίζει αυτό στο προήμιο. Παρότι δεν το λέει με αυτά τα λόγια, η έννοια του δικαιώματος είναι μια πολύ σημαντική έννοια της σύμβασης αυτής. Εξασφαλίζοντας αυτά τα δικαιώματα, θέλει να συνεισφέρει στο να ζούμε ε, σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευμερία. Πέρα από τα ελάχιστα πρότυπα πρόσβαση στην πληροφορία, η συμμετοχή του κοινού τη συμμετοχή, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη μιλάει για πολύ σημαντικές αρχές που αντικατοπτρίζονται και στην ε, εφαρμογή από τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά και στην αναθεώρηση που κάνει η Αρμόδια Επιτροπή. Είναι σημαντικό για να απολαμβάνουμε πραγματικά τα δικαιώματα θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές, διαφανές και συνεπές πλαίσιο στο διεθνές δίκαιο. Και αυτό, ως, ε, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, ισχύει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχει μια ευρύτατη έννοια για το δημόσιο ε, συμφέρον. Ε, επίσης, για την πρόσβαση στην, πληροφορία, στην Δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι έχει ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον, ας πούμε, και να το εξηγήσει. Επίσης, για τις ε, δημόσιες αρχές, τις, εδώ συμπεριλαμβάνει και τις κυβερνήσεις, αλλά και ιδιωτικού φορείς, όταν διενεργούν κάποια καθήκοντα εκ μέρους ε, δημόσιων φορέων και κυβερνήσεων. Καλύπτονται και αυτά από το δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα. Και αυτή η ιδιωτική φορεί, δηλαδή. Έπειτα, η περιβαλλοντική πληροφόρηση είναι αρκετά εκτεταμένη εδώ, θα επανέλθω σε αυτό. Επίσης, απολαμβάνοντα αυτά τα δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία, δίωξη ή παρενόχληση. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκριση λόγω εθνικότητας ε, ή κατοικίας. Ε, εδώ ε, τα κρατικά σύνορα είναι άσχετα για τη συμμετοχή του κοινού. Δεν έχει... Όταν ζητάς, ας πούμε, περιβαλλοντικές πληροφορίες, δεν έχουν σημασία τα σύνορα. Πάμε τώρα στην πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, βασικός πυλώνας το τι είναι περιβαλλοντικό καθορίζει και το πεδίο ουσιαστικά της σύμβασης και τα δικαιώματα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο η κατάσταση του περιβάλλοντος αυτή καθ' αυτή, ε, το νερό, ο αέρας κτλ. αλλά και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, δραστηριότητες, ε, νομοθεσία, ε, δικαστικές αποφάσεις, οικονομικές αναλύσεις, αναλύσεις κόστους-οφέλους που είναι σημαντικές για να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις Όλες αυτές είναι περιβαλλοντικές πληροφορίες. Επίσης, ε, η κατασκευή των κτηρίων, ο σχεδιασμός, ε, πολιτιστικά στοιχεία και αυτά συμπεριλαμβάνονται. Η υποχρέωση των μερών να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση ε, συμπεριλαμβάνουν ένα παθητικό μέρος, έτσι ορίζεται, δεν είναι λιγότερο σημαντικό, δηλαδή τα μέρη ε, είναι αναγκασμένοι να ζητήσουν πληροφορία κατόπιν αιτήματο και θα πρέπει να δίνεται αυτή η πληροφορία το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει και ένα όριο, ένα μήνα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένει ένα μήνα, μπορεί να δώσει πληροφορίε και νωρίτερα. Σε ορισμένε εξαιρετικέ περιπτώσει μπορεί να επεκταθεί αυτή η προθεσμία στου δύο μήνε. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ στην πρόσβαση είναι το τεκμήριο. Μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση μόνο αν σαφώ το συνδέσει με κάποιο λόγο που αναφέρεται. Δηλαδή, εάν η αποκάλυψη αυτή θα επηρεάσει ε, αρνητικά κάποια πράγματα που αναφέρει η σύμβαση. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να ερμηνευθούν με περιοριστικό τρόπο και να λάβουν υπόψη αυτό που αναφέρθηκε στι προηγούμενε παρουσιάσει το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί αυτή η διάδοση, η αποκάλυψη των πληροφοριών. Και για το περιβάλλον, εδώ δεν υπάρχει κανένα περιορισμό Αυτό καθε αυτό για το περιβάλλον. Επίσης, πολύ σημαντικό, είναι κάποιες υποθέσεις που εξετάστηκαν από την Επιτροπή. Η άρνηση θα πρέπει να δοθεί γραπτός ε, και αιτιολογημένη να είναι. Και θα πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις ε, υπάρχουσες διαδικασίες επανεξέτασης. Εάν υπάρχει ε, επιβολή ενός τέλους, θα πρέπει να είναι και αυτό λογικό. Επιβολή τέλους για την πρόσβαση πληροφορίες. Ε, θα πρέπει να είναι λογικό το ποσό και θα πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. Πέρα από αυτές τις παθητικές εντό αγωγικών πληροφορίες, οι δημόσιες αρχές είναι υποχρεωμένε επίσης να εξασφαλίσουν ότι έχουν στα χέρια τους τις απαραίτητες πληροφορίες. Αλλιώς ε, δεν έχει νόημα. Επομένως θα πρέπει να έχουν ε, τις ε, επικαιροποιημένε ε, κατάλληλες περιβαλλοντικές πληροφορίες και να υπάρχει και μια σωστή ροή που θα εξασφαλίσει μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, μέσω μητρών που αφορούν τη μόλυνση και άλλα στοιχεία. Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα στη συμμετοχή του κοινού. Εδώ υπάρχουν ελάχιστα κριτήρια στη σύμβαση για τη συμμετοχή αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να τεθούν ε, τέτοια κριτήρια για παραπάνω από 50 κράτη από το Καζακστάν, ας πούμε, ανατολικά μέχρι το τελευταίο κράτος στη Δύση, ας πούμε, λαμβάνοντας υπόψη τελείως διαφορετικές πολιτικές πραγματικότητε. Ε, το βασικό είναι να έχουμε αυτές τις πληροφορίες ε, πολύ νωρίς, ώστε να έχουμε στη διάθεση μας μια πλειάδα ε, επιλογών θα πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη το αποτέλεσμα της ε, συμμετοχής του κοινού. Αυτό δεν σημαίνει, η συμμετοχή δεν σημαίνει ότι έχεις και βέτο, γιατί συνήθω τα συμφέροντα είναι πολύ ε, διαφορετικά και αντιμαχόμενα, αλλά θα πρέπει όλες οι απόψεις να ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν αντίστοιχες ελάχιστες ε, απαιτήσει με το σχεδιασμό των πολιτικών κτλ. Δεν θα υπήρξαν τις λεπτομέρειες. Και υπάρχουν και γενικοί κανόνες ε, που αφορούν τις κυβερνήσεις κτλ. Πάμε στα τρίτα μέρη. Μιλάμε για την πρόσβαση στις πληροφορίες πάντα. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, ένδικα μέσα ενώπιον δικαστηρίων, αλλά και πιο γρήγορες διαδικασίες. Δυνατότητες επίσης να αμφισβητήσει αποφάσεις ε, για συγκεκριμένες δραστηριότητες και πολύ σημαντικό για άλλες δράσεις δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που παραβιάζουν διατάξεις του, δημοσίου δικαίου, του, διεθνούς δημοσίου, συγγνώμη, του διεθνούς δικαίου που αφορούν το περιβάλλον. Όλες αυτές οι διαδικασίες επιπλέον θα πρέπει να απλούν κάποια ελάχιστα πρότυπα, ισότητα, ε, δικαιοσύνη, ε, να, γίνονται γρήγορα και να μην είναι πολύ δαπανηρές. Γιατί συχνά ε, σε όλα τα κρατη υπάρχουν τέτοιε διαδικασίε, αλλά οι διαδικασίε, ε, α πούμε, οι δικαστικέ είναι τόσο δαπανηρέ που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τι χρησιμοποιήσει κανεί. Α μιλήσουμε τώρα για την Επιτροπή Συμμόρφωση. Εάν. Κοιτάξτε, εδώ σα παρουσιάσω τι απόψει τη ε, Επιτροπή. Εγώ έχω και πιο επικριτικέ απόψει, αλλά δεν έχει νόημα να τι πω εδώ. Ε, τα όσα θα σα παρουσιάσω αφορούν τα πορίσματα τη ίδια Επιτροπή. Από εκεί προέρχονται. Λοιπόν, να σας πω εδώ ότι η Επιτροπή Συμμόρφωσης αναθεωρεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν μπορεί το δικαστήριο να φανταστεί ότι κάποιος εξετάζει δραστηριότητε του, αλλά το κάνει η Επιτροπή ε, Συμμόρφωσης. Και έχει ένα, δώσει ένα μερικό πόρισμα ε, για το δικαστήριο ήδη και σε λίγες εβδομάδες θα το συμπληρώσει αυτό το πόρισμα με ένα συμπληρωματικό. Ε, η Επιτροπή αυτή λαμβάνει ανακοινώσεις υιοθετεί πορίσματα και αυτά τα πορίσματα ε, επικυρώνονται από τα μέρη αργότερα, ε, ούτω ώστε να έχουν ε, ισχύ σε διεθνές επίπεδο. Και παρακολουθεί υποθέσεις όπου κάποια μέρη δεν συμμορφώνονται με κάποιες προϋποθέσεις. Πολύ γρήγορα τώρα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, μέχρι σήμερα υπάρχουν 8 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κατάλογο ε, μερών που δεν έχουν συμμορφωθεί. Αυτή η αναθεώρηση από την Επιτροπή εξαρτάται από τι υποθέσει ε, που φτάνουν στην Επιτροπή. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα κράτη στην πραγματικότητα συμμορφώνονται πολύ λιγότερο από άλλα κράτη-μέλη. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται, απλώ δεν έχει προσφύγει κανένα εναντίον του στην Επιτροπή. Η Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ρουμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Για θέματα που βλέπετε στον κατάλογο για το σημερινό μας θέμα. Σε μία από τις περιπτώσεις, ε, έναντι της Ρουμανίας, η Επιτροπή εξέτασε και τους λόγους άρνησης ε, της ε, παραχώρησης πληροφοριών ε, και το εξέτασε πολύ προσεκτικά. Αυτά είναι τα θέματα που εξετάζει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή για να δει εάν υπάρχει πρόοδος, αν τα μέρη περνούν στη φάση της συμμόρφωσης. Ορισμένα μέρη το κάνουν, είναι πιο προχωρημένα από άλλα και το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύμβαση αφορά όλα τα θεσμικά όργανα και εφαρμόζεται σε όλα τα ε, θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προηγουμένω αναφέρθηκε η τράπεζα. Η, ε, σύμβαση του Άρχους ε, καλύπτει και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά τι περιβαλλοντικέ πληροφορίε. Θα μπορούσαν αυτέ τι πληροφορίε να αφορούν, να αφορούν το δανεισμό κάποιων, την πρόθεση κάποιων project. Η Επιτροπή εξετάζει τι υποθέσει. Η δημόσια πρόσβαση στι πληροφορίε. Ε, η ενωσιακή νομοθεσία ε, που περιορίζει την πρόσβαση ε, στην πληροφόρηση κτλ. Και η πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Όχι μόνο το, πρόσβαση των κρατών μελών, αλλά πρόσβαση στο ίδιο το δικαστήριο για θέματα που αφορούν την ενημέρωση. Η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάστηκε επίση από την Επιτροπή. Είναι πολύ δύσκολο να αποδώσουμε ευθύνε και να τι μοιράσουμε ανάμεσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, γιατί και οι δύο είναι συμβαλλόμενα μέρη. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί νομοθεσία και αυτή η νομοθεσία θα πρέπει να πληρεί κάποια ελάχιστα κριτήρια, ούτω ώστε να γίνεται σεβαστή η σύμβαση άρχου και παρακολουθεί τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τις σωστές επιδόσεις, κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Αυτό που είδαμε ε, για την ενημέρωση και πληροφόρηση ε, είναι οι διατάξεις που λένε ότι οι δημόσιοι φορείς δεν εξηγούν πάντα την άρνησή τους να, να δώσουν πληροφορίες, δεν το κάνουν πάντα εγκαίρως όταν δίνουν τις πληροφορίες. Δεν είναι σαφώς πώς εξορροπούνται τα συμφέροντα ανάμεσα ε, στο, στο, στους λόγους μυστικότητας και στους λόγους αποκάλυψης, ας πούμε, δεν υπάρχει πάντα ισορροπία. Ε, ανησυχίες για την επικοινωνία, εσωτερική ε, επικοινωνία, είναι θέματα που εξετάζει η Επιτροπή Συμμόρφωσης. Λέω, σταματήσω εδώ την παρουσίασή μου. Ε. Ελπίζω ο επόμενος ομιλητής να τα καταφέρει καλύτερα με το PowerPoint. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο δόκτορα Αμπάζη από το κέντρο του Μάστριχτ ε, και το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ για το στην έδρα Ευρωπαϊκού Δικαίου θα μιλήσει για την ισορροπία ανάμεσα στην ε, ε, διαφάνεια και στην εμπιστευτικότητα. Δέκα λεφτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή Αναφορών για την προσοχή σε αυτό το θέμα που καμιά φορά μελείται και σε σχέση με την ε, αύξηση της ε, ε, ευαισθησίας και συνειδητοποίησης. Είναι θετικό το ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία εντάσσονται στην αναθεώρηση και αυτό δείχνει ότι μπορούμε σε σχέση με την επέτειο των 50 ετών τον Ιούλιο να βελτιώσουμε ίσως τα πράγματα σαν συνέχεια αυτών. Θα επικεντρωθώ πράγματι στην ισορροπία μεταξύ της διαφάνειας και του εμπιστευτικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη της διεθνής διαπραγματεύσεις αλλά προτού επισέλθω περισσότερο σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις η νομολογία ή όσον αφορά μια ισόρροπη παρουσίαση, θέλω να τονίσω τη διαφοροποίηση που καμιά φορά ξεχνάμε μεταξύ δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες και κοινοβουλευτικής, ε, κοινοβουλευτικού χαρακτήρα πρόσβασης ε, σε πληροφορίες. Καμιά φορά ξεχνάμε αυτή τη διαφοροποίηση, μια και πολλές φορές οι ίδιοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι βρίσκονται σε νομική κατάσταση όπου έχουν ε, σε σχέση με την αναφορά στον κανονισμό 1049 για την πρόσβαση σε πληροφορία, το πιο σημαντικό στοιχείο για αυτή τη διαφοροποίηση είναι ότι η δημόσια πρόσβαση είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες και έτσι γίνεται δημόσιο αγαθό η πρόσβαση αυτή ενώ η άλλη αφορά το πρωτογενές δίκαιο και σε σχέση με το άρθρο 219 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζεται περαιτέρω στους εσωτερικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε σχέση και με τις ρυθμίσεις της Διοργανικής Συμφωνίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο όπου υπάρχουν περισσότερο εξειδικευμένες ε, ε, ρυθμίσεις το πιο συγκεκριμένο για αυτή τη συγκεκριμένη πρόσβαση είναι ότι είναι προνομιακού χαρακτήρα. Δηλαδή δεν, δεν γίνονται δημόσιες οι πληροφορίες, δεν αποκτούν δημόσιο καθεστώς. Και παρόλη την, την βελτίωση σε σχέση με την κοινοβουλευτική πρόσβαση θα πρέπει να δούμε κατά πόσον βελτιώνεται η γενική πρόσβαση όσον αφορά τα θέματα ε, εμπιστευτικότητας και διαφάνειας. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και προαναφέρθηκε ότι υπάρχει κάποια ανάγκη εμπιστευτικότητας, υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, διαπραγμάτευσης ε, όπου υπάρχει ένα αναγκαίο επίπεδο, ε, ελάχιστο επίπεδο εμπιστευτικού χαρακτήρα. Τονίζω όμως, καθώς αυτό είναι αναγκαίο, βλέποντας σε σχέση με το διεθνές πλαίσιο στην πρακτική εφαρμογή το τι συμβαίνει θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει μια ολόκληρη σειρά περιπτώσεων προσφυγών στο 10 Βλέπουμε και τα επιχειρήματα της Επιτροπής και του Συμβουλίου που επεκτείνουν αυτή την λογική αναγκαστικού χαρακτήρα ή έκτακτου χαρακτήρα με ευρύτερα πλαίσια όσον αφορά την κάλυψη της εμπιστευτικότητας. Είναι όμως σημαντικό να τονίσουμε ότι πρόσφατα είδαμε αρκετά σημαντικά νέα νομικά όρια σε σχέση με το αποδεκτό επίπεδο εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα αξίζει να αναφέρουμε την περίπτωση ε, ε, που, ε, προσφυγής που ασκήθηκε κατά του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση σε στοιχεία πληροφόρησης ε, όσον αφορά διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αυτό σε σχέση με συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, είναι η πρώτη περίπτωση όπου το 10 συγκεκριμένα ζήτησε από το Συμβούλιο να αποδείξει ότι η γνωστοποίηση αυτών των στοιχείων ουσιαστικά και πράγματι θα υπονόμευε τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Σε σχέση λοιπόν με το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας θα μπορούσε λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να εξεταστεί το θέμα της εμπιστευτικότητας. Ενώ σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν δέχεται ευρύτερες απαιτήσει ε, το δικαστήριο όσον αφορά αυτή την εφαρμογή της διακριτικής ευχέρειας και ζητεί να αποδειχθεί η επιζήμια επίπτωση σε σχέση με τη δημοσιοποίηση στις δημόσιες αυτές διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε ότι το περιθώριο σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να είναι συμφωνία για την μετάθεση, μεταφορά χρηματοοικονομικών στοιχείων όσον αφορά για παράδειγμα την καταπολέμηση και πρόληψη της τρομοκρατίας τονίζεται ο συνταγματικός χαρακτήρας από το δικαστήριο μέσα στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων ότι κάποιες από αυτές τις διατάξεις και είναι πολύ σημαντικό το ότι αθίγονται θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και η μεγαλύτερη εξειδίκευση στο πλαίσιο αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν γίνεται δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ισχυρίζονται και να επικαλούνται ευρύτερη, ε, ε, ευρύτερη αρμοδιότητα όσον αφορά την άσκηση διακριτικής ευχέρειας για την εμπιστευτικότητα από πλευράς τους. Αυτό το οποίο βλέπουμε διαρκώς και συστηματικά τι είναι και ίσως και όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων αλλά επίσης και σε άλλες περιπτώσεις είναι ότι η λογική υπέρ της εμπιστευτικότητας που λειτουργεί είναι για να υπάρχει λέει εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσόμενων εταίρων έναντι ε, της ε, ε, εμπιστοσύνης σε σχέση με ένα ευρύτερο πλαίσιο για τους πολίτες ανοίγοντας αυτά τα έγγραφα σε δημόσια πρόσβαση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπόκει χρησιμοποιούνται αυτά τα επιχειρήματα σε σχέση με την εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσόμενων που έχει προτεραιότητα έναντι της διαφάνειας και του πνεύματος εμπιστοσύνης, κλίματος εμπιστοσύνης υπέρ των πολιτών. Και βλέπουμε <clears throat> ότι αυτό είναι ένα θετικό παράδειγμα σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν. Είναι μία από ολόκληρη σειρά συμφωνιών όπου το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι υπέρ του ότι πρέπει να αποκατασταθεί, να διασφαλιστεί το, πνεύμα, το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσόμενων, συμβαλόμενων εταίρων. Είναι σημαντικό εδώ να δούμε τα νομικά όρια τα οποία αναπτύσσονται και εκπονούνται. Απ' την άλλη πλευρά να δούμε τη λογική και το πνεύμα υπέρ της εμπιστευτικότητας που εξακολουθεί να είναι συστηματικού χαρακτήρα από πλευρά της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Και οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων TTIP είναι κάτι το οποίο αποκαλύπτει πολλά πράγματα σε σχέση με τις, με τις διαδικασίες αυτές. Σε σχέση τώρα με την, ε, το κοινοβουλευτικό πλαίσιο είναι ένας άλλος τομέας όπου μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα όπως προανέφερα το δικαίωμα σε κοινοβουλευτική πρόσβαση είναι συνταγματικού χαρακτήρα, όμως εξειδικεύεται περισσότερο από εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς ε, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και <clears throat> διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας που έχει το Ευρωκοινοβούλιο με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές οι συμφωνίες συζητήθηκαν και αυτές και κλεισμένων των θυρών κατά το παρελθόν και δεν είναι υποχρεωτικά υπέρ της, ε, του ανοίγματο του πλαισίου ε, αυτών των πληροφοριακών στοιχείων ε, διότι βλέπουμε ότι η πρόσβαση σε τέτοια έγγραφα και κλεισμένων των θυρών αν δεν μπορούν να γίνουν σημειώσεις να υπάρξουν φωτοαντίγραφα τότε εδώ υπάρχει περιορισμός των δικαιωμάτων και των διαδικασιών. Ενώ βλέπουμε ότι η πρόσβαση βελτιώνεται όσον αφορά την προώθησή της βλέπουμε ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά ότι διαγράφεται ο κίνδυνος αυτό να αποβαίνει εις βάρος της ικανότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημόσια να συζητήσει αυτά τα θέματα με βάση αυτά τα στοιχεία, με βάση στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται και κλεισμένων των θυρών στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Υπάρχουν εδώ θέματα τα οποία αφορούν πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη συμφωνία Σαντάνια και όπου θεωρούμε ότι η διασφάλιση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρόσβαση σε πληροφορίες και στην περίπτωση της προηγούμενης εβδομάδας εδώ από πλευράς του δικαστηρίου αναφέρθηκε ότι εννέα ημέρες η αποστολή εγγράφου ε, και όχι άμεσα όπως απαιτείται από τη συνθήκη είναι υπερβολική καθυστέρηση και ότι εδώ πράγματι έχει το δικαίωμα άμεσα και σε όλες τις φάσεις να ενημερώνεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα αυτά τα στοιχεία. Τονίζει λοιπόν το δικαστήριο σε αυτήν την περίπτωση το πλήρες φάσμα, το πλήρες εύρος της ανάγκης εφαρμογής αυτών των διατάξεων για πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνει και να διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο. Στην πρακτική εφαρμογή υπάρχει όμως κάποια σύγχυση, δηλαδή ποιος θα είναι ο αποδέκτης ή τι θα συμβαίνει σε σχέση με τη ε, διαδικασία αυτή για το άνοιγμα πληροφοριών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε, επειδή δεν βρίσκονται όλα τα θεσμικά όργανα ε, σε ίσο βαθμό στην ίδια πλευρά και βλέπουμε ότι ενώ η Επιτροπή έχει σε κάποια σημεία ενδώσει, το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να υποχωρήσει. Και για την πρόσφατη συμφωνία Σαλδάνια, για παράδειγμα, δεν διαβιβάστηκαν πληροφορίες έγκαιρα στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι υπήρξαν σημαντικές νομικές εξελίξεις και όσον αφορά την ομολογία και όσον αφορά την δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά και την κοινοβουλευτική πρόσβαση αλλά συμφωνώ σε σχέση με τα συμπεράσματα ότι πρέπει να γίνει μια πιο ανοιχτού χαρακτήρα συζήτηση για το θέμα της εμπιστευτικότητας για το πώς δηλαδή απόρριτα ε, θέματα τα διαχειριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προστατεύουμε. Είναι σημαντικό να γίνει αυτή τη χρονική στιγμή μια συζήτηση για το πώς δηλαδή η ισορροπία αυτή διασφαλίζεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ εμπιστευτικότητας και δημόσιου χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και νομίζω και ενθαρρυντικά για εμάς που ζητάμε συνέχεια να σταματήσουν οι συναντήσεις και κλεισμένων των θυρών. Ε, και μάλιστα ε, ε, οι δικές μας συνεδριάσεις μαγνητοσκοπούνται και χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν αυτά που κάνουμε. Ενώ άλλε επιτροπές έχουν την τάση κάποια κομμάτια της συνεδρίασης να τα διεξάγουν και κλεισμένων των, ειδών, των θυρών. Συγγνώμη. Είμαι περήφανη λοιπόν που είμαι μέλος ετούτης της Επιτροπής. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους ή Μακρέτε Άουκεν. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους, προσκεκλισμέ... τους προσκεκλημένους μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, παλιά σύμβαση, διότι είναι οικογενειακό μας μωρό, διότι ο αδερφός μου ήταν τότε ε, υπουργός ε, περιβάλλοντος και ήταν ε, ο εμπνευστής ε, της ε, πρώτης σύμβασης του Όρχους. Νομίζω όμως ότι δεν είναι μόνο θέμα νομικών αγώνων, είναι και πολιτικοί αγώνες που παλεύουμε εδώ στην Δανία. Έχουμε μόνιμο πόλεμο για το θέμα της διαφάνειας. Κατά τη θητεία μου στο Δανέζικο Κοινοβούλιο, αλλά και εδώ, διαπιστώνω ότι κάθε φορά που οι θεσμοί έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις πόρτες, τις κλείνουν. Αυτό πιθανότατα να μην ισχύει στη, Δανία, στη Σουηδία, στη Δανία όμως σίγουρα ισχύει. Και συχνά είναι τρομερό να ακούει κανείς έναν επίτροπο ή έναν υψηλό αξιωματούχο εντός της Επιτροπής να λέει ότι ο στόχος είναι να προστατευτούν οι αξιωματούχοι οι υπάλληλοι. Διότι είναι ένας ε, σύμβουλος ε, θα πρέπει να μπορεί να κάνει και λάθη, αλλά μερικά λάθη σκοτώνουν όλους και δεν έχουν καταλάβει ότι ο καλύτερος τρόπος να έχουμε καλούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους ε, είναι να υπάρχει διαφάνεια και σεβασμός για τα πρόσωπά τους. ακόμα και μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας ε, και μετά τον ε, χάρτη, ζητήσαμε κάποιοι εδώ στο Κοινοβούλιο την αναθεώρηση του 1049. Μας προειδοποίησαν όμως διότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο ήταν κατά. Δηλαδή αν ξανανοίγαμε το κουτί ε, θα ήταν χειρότερη η κατάσταση από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή και είδαμε πρωτοβουλίες από πλευράς της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποδυνάμωση του 1049, κάτι που μας βάζει σε πολύ δύσκολη θέση. Δυσκολεύαμε να δω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε Εάν δεν υπάρχει πραγματική βούληση εντός του Συμβουλίου και της Κομισιόν να πληρούν τις υποχρεώσεις τους για σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου. Και το μόνο σημείο όπου έχω μια μικρή επιφύλαξη είναι η σε διάλογοι. Ε, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια μετά, αλλά ξέρετε πόσο ευάλωτο είναι το κοινοβούλιο στο lobbying. Εάν λοιπόν τα άλλα θεσμικά όργανα έχουν πλήρη διαφάνεια κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων, θα περιθωριοποιηθούμε ακόμα περισσότερο στην διαδικασία. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός αυτό. Όσοι διστάζουν γνωρίζουν το παιχνίδι. Εν μέσω λοιπόν μιας ε, διαδικασίας διαπραγμάτευσης ε, και αυτό είναι το θέμα των τρίμερων διαλόγων. Και μπορούμε να δημοσιεύσουμε όλα τα στοιχεία εκ των υστέρων, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε πόσο αποδυναμώνεται την θέση του Κοινοβουλίου εφόσον ε, δεν ε, υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσει από το Συμβούλιο. Και ναι, το ξέρω, λυπάμαι που το λέω, αλλά εκείνοι έχουν ε, τα χρήματα. Ε, ε, οι, οι μεγάλοι λομπίστες εννοώ, έχουν όλα τα όπλα στη διάθεσή τους. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Ελεονόρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δημόσια κρόαση και πολύ ενδιαφέρουσα οι παρουσιάσεις. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα για ένα ουσιαστικό θέμα που συνδέεται άρρηκτα με τα όσα ακούσαμε σήμερα το πρωί και αφορά την τη διαφάνεια και την πρόσβαση στις πληροφορίες σε σχέση με τα μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται στην Ευρώπη. Και πιο συγκεκριμένα, αυτά που έχουν ένα χαρακτήρα και μία διάσταση διασυνοριακή. Και όπου εμπλέκονται δηλαδή πάνω από ένα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την ε, ιστορία που επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια για το ΤΑΒ, για το έργο τρένου υψηλής ταχύτητας το Ρήνου Λιών, που είναι ένα έργο το οποίο αντιμετώπισε μεγάλες αντιστάσεις ε, βάσει επιχειρημάτων πάντα. Το, το αντιπιχείρημα στην κατασκευή του ήταν ότι είναι τι αυτή η σιδηροδρομική γραμμή. Υπάρχει ούτως ή μια σύνδεση σιδηροδρομική που έχει ανακαινιστεί ανάμεσα στις δύο πόλεις και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη και λόγος να φτιάξουμε ένα, μια νέα σιδηροδρομική γραμμή ψηλής ταχύτητας δεν υπάρχει επαρκής ροή ούτε επιβατών ούτε εμπορευμάτων οι κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να ακουστεί η φωνή τους. Ένας από τους φορείς που δημιουργήθηκε για να ακούσει τη φωνή των πολιτών είναι ένα είδος παρατηρητηρίου όπου συμμετέχουν οι διάφορες τοπικές ε, αρχές, διάφοροι δήμαρχοι κτλ. Φτιάχτηκε με έναν πολύ αδέξιο τρόπο, πολύ άκομψο, απότομο θα έλεγα. Φημώθηκαν εντελώς οι ενάντιες φωνές και σε αυτό το παρατηρητήριο εδρεύουν μόνο και αποκλειστικά οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων και δήμων που είναι υπέρ ε, τις οργανωτικές που είναι οι, οι δήμοι και που αποφελούνται ουσιαστικά από αυτή την ε, γραμμή. Θα θέλαμε να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών της περιοχής αυτής, των κατοίκων της περιοχής αυτής. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και συμμετοχή και πρόσβαση στην τεκμηρίωση ούτως ώστε η περιβαλλοντική νομοθεσία να μπορεί να εφαρμοστεί σωστά. Σε ποιο βαθμό η Ευρώπη γνωρίζει τέτοιες συγκεκριμένες καταστάσεις που δεν συμβαίνουν μόνο σε μία χώρα ή σε μία πόλη, αλλά μιλάμε για διασυνοριακά έργα τα οποία αφορούν πολλά κράτη και πόλεις και που υπάρχουν πολλές απόψεις που δεν ακούγονται όμως. Εδώ έχουμε το πολύ ισχυρό εθνικό επίπεδο που ακούγεται τη φωνή του, αλλά τα υπόλοιπα επίπεδα, οι υπόλοιποι φορείς, οι κάτοικοι κτλ. πώς θα ακουστούν, πώς εξασφαλίζεται την συμμετοχή ε, και την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και πώς είναι δυνατόν να βελτιωθεί αυτή η πτυχή στο μέλλον, ούτω ώστε να ακουστεί περισσότερο η φωνή των πολιτών ε, που θέλουν να εκφραστούν για τέτοια θέματα που αφορούν έργα υποδομής τεράστια, που δεν ωφελούν όμως τις περιοχές αυτές, αλλά που πληρώνονται αντίθετα ε, από τις τσέπες των πολιτών αλλά και των μελλοντικών γενιών και έχουν και μια αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι και εμείς πληρώνουμε αλλά και οι επόμενες γενιές θα πληρώσουν για έργα τα οποία είναι λάθος, ε, είναι λάθος επιλογές και δεν έπρεπε να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Μαγκρέτε, σύντομη παρατήρηση. Ναι, όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ήμουν σκιώδης εισηγήτρια για την εφαρμογή της παλαιάς συνθήκης στο Κοινοβούλιο. Και θεωρούσα ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε την ε, παλαιά ε, σύμβαση. Αλλά υπήρχε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, παρότι στήριζαν το υπόλοιπο της σύμβασης που ήταν κατά της ε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πράγμα που σημαίνει ότι κατά την νομοθετική διαδικασία στο Κοινοβούλιο ε, το θέμα αυτό ε, εμποδίστηκε από μια πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν δύσκολο για μένα να καταλάβω πώς ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν τηρούμε τη συνθήκη. Το δικαστήριο θα έπρεπε κανονικά να είναι ο φορέα που το χειρίζεται αυτό, αλλά πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση, διότι δεν είναι πολύ εύκολο, σας το λέω ειλικρινά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας δώσω τη δυνατότητα να απαντήσετε στις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Ε, δεν σας έθεσαν ακριβώς ερωτήσεις, ε, αλλά να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω. Εγώ θα κάνω κάποιε παρατηρήσεις και νομίζω μετά θα θέλει και η καθηγήτρια Λάινο να πάρει το λόγο. Αναφέρθηκε ο πόλεμος που γίνεται όχι μόνο στη Δανία αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είναι κάπως υπόγειος, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει. Μέρος του προβλήματος είναι αφενός η αναθεώρηση της νομοθεσίας, ε, από την άλλη έχουμε το τι γίνεται στην πράξη. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί το δίκαιο ώστε να μπορεί κανείς να χειρίζεται προβλήματα στην πράξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί έτσι να εξαλείψει κανείς όλα τα προβλήματα, πάντα θα υπάρχει αντίσταση, διαφωνούντες ε, κλπ. Αλλά αυτή είναι η φύση της πολιτικής. Ιδιαίτερα προβληματικό όμως στην παρούσα κατάσταση είναι το εξή. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και η Κομισιόν μόνο έχει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας. Στην πράξη όμως βλέπουμε και το αναφέρουμε αυτό ρητά στην έκθεσή μας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρότι η νέα Επιτροπή φέρεται να έχει θέσει ως προτεραιότητα την διαφάνεια, τουλάχιστον αυτό έκανε όταν ανέλαβε καθήκοντα, εάν δούμε τις εξηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε δικαστικές υποθέσεις, αγωνίζεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και να υπάρχει ε, να ισχύει η εμπιστευτικότητα αυτομάτως ε, αντί να ισχύει η διαφάνεια αυτομάτως και να υπάρχουν εξαιρέσεις από αυτήν. Μήπως θα, θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, πιο γενικός, ανοιχτός, δημοκρατικός διάλογος πάνω στα θέματα αυτά. Αυτό ακριβώς θέλουμε να προτείνουμε μία συγκεκριμένη πρόταση της εκθεσής μας μπορεί να χάθηκε λίγο ε, μεταξύ των άλλων, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την διοικητική διαδικασία έχει υποβάλει ένα μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιστέκεται σε αυτό, λέει ότι δεν απαραίτητο κάτι τέτοιο. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να μην έχει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας επισήμως, άτυπα όμως προωθεί έτσι τη συζήτηση. Νομίζουμε ότι αυτό θα ήταν καλή ιδέα να γίνει. Επίσης, ε, κάτι που δεν συζητηθήκε πολύ ούτε εδώ σήμερα και μπορεί να μην είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος, ε, αλλά θεωρούμε ότι ε, η διαβάθμιση των εγγράφων και δεν αναφέρομαι μόνο στα στα έγγραφα με υψηλή διαβάθμιση εμπιστευτικότητας θα πρέπει να γίνει συζήτηση ανάμεσα στη σχέση των κανόνων για την πρόσβαση στα έγγραφα και των κανόνων για την εμπιστευτικότητα. Και έχουμε προχωρήσει πολύ σε σχέση με το 2001 όταν ε, υιοθετήθηκε ο κανονισμός. Ε, θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τη σχέση αυτών των δύο. Μάλιστα ήδη πριν χρόνια πρότεινα ότι θα πρέπει να υπάρχει νόμος περί εμπιστευτικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα πρέπει να καθοριστούν τα επίπεδα αλλά και τα όρια της εμπιστευτικότητας. Και τέλος, όσον αφορά τον τριμερή διάλογο, είναι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι θα προτείναμε ποτέ μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποκαλύπτει τις ε, διαπραγματεύσεις ε, το πρόβλημα όμως ε, είναι ότι η διαδικασία αυτή μοιάζει με διπλωματική διαπραγμάτευση ε, μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και μπορεί κανείς ε, να αμφισβητήσει τη χρησιμότητα ενός τέτοιου μέτρου σε μια δημοκρατική διαδικασία. Αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο, διότι η λύση, μπορεί, η λύση πρέπει απαραίτητα να είναι διαθεσμική. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί, κάπου όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η καθηγήτρια Κέρτσιν. Ε, το λόγο έχει η καθηγήτρια Λέινο Σάντερ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση, με την αναθεώρηση του κανονισμού. Νομίζω ότι θα είναι μια πολλά υποσχόμενη διαδικασία και κατόπιν θέλω να αναφερθώ στους τριμερείς διαλόγους όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού. Είχα ασχοληθεί με την διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση του 1049. Καταλαβαίνω ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν ανοίξουμε τη διαδικασία αυτή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μειονότητα που μπορεί να μπλοκ ψηφία που να μπορεί να πλοκάρει την κατάσταση στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι σίγουρα εναντίον της ε, διεύρυνσης της διαφάνειας. Πολύ θετική νομολογία ε, έχουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την πρόσβαση στα έγγραφα. Σε περίπτωση που το έχουμε αυτό ε, θα μπορέσουμε να περάσουμε μια τέτοια πρόταση. Αλλά υπάρχει κίνδυνος αν ανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά όμως τα διοικητικά θέματα που επίσης είναι θέμα που θίξαμε, χρειαζόμαστε νομοθετική επέμβαση, διότι βλέπουμε πολλούς να ξεφεύγουν ε, λόγω του καθεστώτος ε, μυστικότητας που υπάρχει. Το δικαστήριο έχει στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να βρούμε υπόθεση όπου δεν έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά που ήθελε από το δικαστήριο. Ο μόνος τρόπος ε, να αλλάξουμε το καθεστώς ε, είναι ο, ο νομοθετικός. Όσον αφορά λοιπόν ε, τις ε, υποθέσεις επιπαραβάση, πρόκειται για νομοθετικές διαδικασίες, παρότι δεν εμπίπτουν αυστηρά στην νομοθετική διαδικασία. Είναι λοιπόν θέματα όπου όπως είπα και πριν υπάρχει ο κίνδυνος ε, να περιορίσουμε τα ε, εθνικά συστήματα διαφάνειας. Είναι λοιπόν προβληματική η κατάσταση. Επίσης υπάρχουν τομείς όπου υπάρχουν δυνατότητες, ε, για παράδειγμα στις διεθνείς σχέσεις. Μπορούμε με ερμηνεία ή με την εξέβρεση νέων πρακτικών χωρίς να αλλάξουμε το ρόλο, ε, να αλλάξουμε την κατάσταση και η διαμεσολαβήτρια έχει βοηθήσει πολύ στην προσπάθεια αυτή. Το άλλο θέμα το οποίο θέλω να αναφέρω είναι η τριμερής διάλογη. Έχω δει την κατάσταση και από πλευρά του Συμβουλίου. Και μία από τις μεγάλες νίκες μας ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας ήταν οι ανοιχτές συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι οι νομοθετικές συμφωνίες συνάπτονται όλο και περισσότερο σε ε, επίπεδο κορεπέρ. Δεν φτάνουν ποτέ στο Συμβούλιο και ένας από τους λόγους είναι ότι όλοι γνωρίζουν ότι τα Συμβούλια Υπουργών είναι ανοιχτών ενώ η κορεπέρ δεν είναι. Και σε κάποιο βαθμό καταλαβαίνω ότι τα κράτη-μέλη χρειάζονται κάποιον χώρο εμπιστευτικότητας όπου πρέπει να μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες ε, χωρίς ε, να χάνουν ε, το γοητρό της την αξιοπιστία τους δεν θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε ποτέ τελείως από αυτό. Ταυτόχρονα αποτελεί πρόβλημα ότι το πιο αποφασιστικό τμήμα της νομοθετικής διαδικασίας είναι απολύτως κλειστό. Αυτό είναι πρόβλημα και για τα εθνικά κοινοβούλια, διότι δεν γνωρίζει τις θέσεις του Συμβουλίου, δεν ξέρει πώς έχουν εξελιχθεί οι τριμερείς διάλογοι και δυσκολεύονται πολύ να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις σε πραγματικό χρόνο κάτι που δημιουργεί και ένα πρόβλημα νομιμότητας για το Συμβούλιο, διότι και τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να υπάρχει πολιτική συζήτηση σχετικά με τα όρια της εμπιστευτικότητας σε συνομοθετική διαδικασία, διότι αυτή τη στιγμή τα όρια αυτά έχουν καθοριστεί με βάση μονομένα αιτήματα και από πλευράς του Συμβουλίου βλέπουμε μια επιχειρηματολογία που ουσιαστικά κατηγορεί τους πολίτες που ε, διαταράσσουν την νομοθετική διαδικασία. Ε, αυτό όμως είναι παραβίαση του δικαιώματος των πολιτών να συμμετέχουν. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και όχι μετά την σύναψη των συμφωνιών. Θα πρέπει έτσι λοιπόν να καθορίσουμε τον χώρο για πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο με πραγματικό δικαίωμα συμμετοχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστώ κύριε καθηγήτρια. Παρακαλώ καθηγήτης Έμπεσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σχολιάσω αν επιτρέπετε δύο θέματα που αναφέρθηκαν από προλαλήσαντες. Το πρώτο για τα σχέδια υποδομών και φυσικά αυτά τα σχέδια υποδομών αναφέρουν αυτό το θέμα για το θέμα των πληροφοριών μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το να έχει κανείς πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα στοιχεία για προγράμματα ή σχέδια υποδομών είναι σημαντικό για τη συμμετοχή του δημοσίου, διότι χωρίς αυτή η πρόσβαση στη σωστή πληροφόρηση δεν μπορεί κανείς να συμμετάσχει εύθετα και είναι ένα θέμα επιδόσεων σε σχέση με τη συμμετοχή, αλλά είναι και ένα θέμα ακόμα και χωρίς ε, συγκεκριμένη αφορά στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων. Εδώ σε σχέση με αυτή τη σύμβαση έχουμε κάποια πείρα σε σχέση με θέματα συμμόρφωσης όσον αφορά τα, τις υποδομές για τα ανανεώσιμα και σε σχέση με τις μεγάλες διασυνδέσεις όσον αφορά αιωλική ενέργεια, τις ανεμογεννήτριες και είναι λοιπόν σημαντικό και μπορεί να γίνει και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όλα τα θεσμικά όργανα σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, Ιταλία, Γαλλία, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινοτικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα δημόσιων αρχών πρέπει να ισχύει αυτό. Ισχύει επίσης και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά θέματα περιβαλλοντικά και βλέπουμε ότι πολύ λίγες πληροφορίες δεν θα, θα μπορούσαν να εξαιρούνται. Όταν έχουμε θέματα, για παράδειγμα, δημόσιων προσφορών, που ίσως κάποια θέματα πρέπει να είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, όλα τα άλλα πρέπει να δημοσιοποιούνται πρέπει να δημοσιοποιούνται αρκετά πρώιμα, αρκετά νωρί, ώστε το κοινό να μπορεί να συμμετέχει για όλε τι εναλλακτικέ δυνατότητε. Και όπω τόνισα, κατά τη διάρκεια τη διαδικασία λήψη απόφαση πρέπει να γίνεται αυτό και όχι μεταγενέστερα με καθυστέρηση, για να μπορεί κανεί να δει τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και να εφαρμοστεί. Απέτηση σε σχέση με την Επιτροπή για θέματα συμμόρφωσης είναι ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να ε, ε, αποτελούν αντικείμενο συμμόρφωσης και στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε σε όλες τις δυνατότητες να υλοποιούνται. Πρέπει να δούμε σε σχέση με την σύμβαση όρχους ότι όλα αυτά τα στοιχεία έχουν τη δική τους σπουδαιότητα. Πρόσβαση, προσπερασμότητα σε θέματα δικαιοσύνης. Και βλέπουμε ότι σε σχέση με αυτό ότι σε πολλές εθνικές νομοθεσίες γίνονται, ε, πρέπει, πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Δεν έχουν γίνει οι αλλαγές σε σχέση με την ε, επικαιροποίηση στα κράτη-μέλη όσο όφυλαν και στη Σουηδία από την οποία προέρχομαι σωστά διαπιστώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν ήταν παραβίαση της νέας συνθήκης αλλά το δικαστήριο είπε ότι η Σουηδική νομολογία δεν συμμορφωνόταν με τις διατάξεις και προδιαγραφές της Σύμβασης του Όρχους. Και όταν κάνουμε λόγο για την εφαρμογή των διατάξεων Όρχους στα κράτη-μέλη, Όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γενικά ήταν σε μεγάλο βαθμό υπέρ της προαγωγής ε, της ε, ε, ορθής εκτέλεσης αυτών των προδιαγραφών για την ε, προσπελασιμότητα. Αναφέρομαι τώρα στο θέμα το ότι υφίσταται ένα ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκεκριμένες ε, προδιαγραφές για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Νομίζω το 2002-2003 πολύ αρκετά νωρίς έγινε πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ε, νομοθεσία για την ε, συμμετοχή στις ε, διαδικασίες για το δημόσιο χαρακτήρα δεν προήχθησαν αυτά όπως έπρεπε και γι' αυτό εξακολουθεί να είναι ένα θέμα επί του οποίου την, προσπαθεί να ασκεί στην επιρροή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δούμε σε σχέση με την συμμόρφωση ότι υπήρξε ένα παράπονο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υιοθέτησε αυτή την νομοθεσία και αυτό θα σήμαινε μη συμμόρφωση. Αυτό όμως το οποίο θα μπορούσα εγώ να αναφέρω είναι ότι ενώ νομοθεσία υιοθετήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ε, υλοποίηση από πλευρά των κρατών ε, μελών ε, και τη σύμβαση του Όρχους όσον αφορά την συμμετοχή του κοινού σε αυτές τις ανοιχτές διαδικασίες η προαγωγή σε σχέση με θέματα δικαιοσύνης από πλευρά του δικαστηρίου πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία για τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία πολύ σωστά απαντήθηκαν. Εγώ θα επιστρέψω σε ευρύτερα θέματα τα οποία όταν επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε λεπτομέρειες ή σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, ξεχνάμε γιατί ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Γιατί είναι σημαντική διαφάνεια, γιατί ενδιαφερόμαστε, γιατί θέλουμε να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρακτική εφαρμογή όσον αφορά την ε, δημιουργία υποψίας ή ενός κλίματος ε, απουσίας εμπιστοσύνης ε, όταν βλέπουμε ότι παρακρατούνται πληροφορίες από θεσμικά όργανα και οι πολίτες παραμένουν εκτός και αποξενώνονται. Έχει τεράστια υπαρξιακή σημασία αυτό το θέμα για τους πολίτες. Είναι, ας το πω έτσι, συγκολητική ύλη που δημιουργεί την επαφή μεταξύ των πολιτών, του, της υποδομής δηλαδή, των θεμελίων και του επικοδομήματος. Ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, τα θέματα εμπιστευτικού χαρακτήρα στους τριμερείς διαλόγους, οι διεθνείς συμβάσεις, ε, όλοι αναγνωρίζουμε είτε είμαστε πανεπιστημιακοί είτε όχι ότι υπάρχει ανάγκη μεν να διασφαλίζεται αυτή η εμπιστευτικότητα. Όμως από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να δημιουργείται ένας ε, φόρτος, μια κόποση όσον αφορά τα θέματα διαφάνειας και να τα αφήνουμε χωρίς να προάγονται. Είναι τεράστια σημασία διότι και πάλι θα επανέλθω στις διαπραγματεύσεις ως παράδειγμα για την TTIP. Δημιουργούνται τόσες απογοητεύσεις ή τέτοια απογοήτευση στους πολίτες ότι ουσιαστικά ο χαρακτήρας αυτός μπορεί να υπονομεύσει τις ίδιες τις διαπραγματεύσεις στην έκβασή τους με αυτή την αρνητική τοποθέτηση. Είναι θεμελιώδης σημασίας λοιπόν τα θέματα εμπιστοσύνη. Και αυτές είναι οι σημαντικές διαστάσεις σε θέματα ισορροπίας που πρέπει να θυμόμαστε όταν λέμε ότι υπάρχει ανάγκη να επανεξετάσουμε τα θέματα αυτά και γιατί ακριβώς είναι τόσο σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σημαντικά θέματα που τονίσατε ορισμένοι μίλησαν για τις διαφορές ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και στην έλλειψή της. Από εκεί που να ξεκινήσουμε. Ε, στην Ευρώπη σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ακραία παραδείγματα δυσπιστίας και έλλειψης εμπιστοσύνης γενικά. Ε, θα πρέπει να συζητήσουμε τι σημαίνει εμπιστοσύνη και να μην, και να ε, τροφοδοτούμε αυτό το φαύλο κύκλο δυσπιστίας. Ε, η εμπιστοσύνη πρέπει να ενισχυθεί. Και αυτό είναι που είναι σε κρίση σήμερα στην Ευρώπη, η έλλειψη εμπιστοσύνη. Κλείνω λοιπόν το πρώτο τμήμα της ακρόασή μα και δίνω το λόγο τώρα στην Γιούλια Πιτέρα, που θα είναι πρόεδρος του δεύτερου πάνελ. Ελπίζω αργότερα να ξανάρθω στην συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλή συζήτηση. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Θα προεδρεύσω σε αυτό το δεύτερο πάνελ και το θέμα του είναι η ελευθερία της ενημέρωσης στην πράξη. Ποιος είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή, τι κάνει η κοινωνία των πολιτών και θα ακούσουμε επίσης τι έκανε και η τελευταία Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το τρίτο θέμα μας, ε, η Ολλανδική Προεδρία. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Φάρ Ρίγκαν, που είναι ο τμήματάρχης του, τμήματος, ε, του ερευνητικού συντονιστικού τμήματος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και θα μιλήσει για την δυνατότητα πρόσβασης του κοινού ε, σε πρόσφατες έρευνες. Πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες εννοώ Καταρχάς, ευχαριστή, εκ μέρους της κυρίας προς την Επιτροπή Αναφορών και προς το Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε κάποιες από τις απόψεις μας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Αυτή η πλατφόρμα συζήτησης που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ζωτική σημασία για τη δραστηριότητα του διαμεσολαβητή και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Πριν πω σε συγκεκριμένα μου θέματα, θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στα τελευταία σχόλια της κυρίας Βίκστρομ. Την κρίση εμπιστοσύνη που έχουμε στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στα θεσμικά τη όργανα. Και θα πρέπει να οικοδομηθεί στο μυαλό και στην καρδιά των Ευρωπαίων πολιτών αυτή η εμπιστοσύνη. Μαζί με την εμπιστοσύνη έρχεται και η νομιμότητα και πιο αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διαφάνεια είναι σημαντική για να υπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη. Ο διαμεσολαβητής παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ε, το ρόλο αυτό τον δίνουν οι συνθήκες, να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στου πολίτε και στην Ένωση και στα θεσμικά τη όργανα. Και υπ' αυτή την έννοια, δεδομένης τη σημασία της διαφάνεια είναι λογικό που η διαφάνεια βρίσκεται πάνω-πάνω στην ατζέντα του διαμεσολαβητή. Και αυτό απεικονίζεται και στο γεγονός ότι πάνω από το 30% των δικών μας ερευνών κάθε χρόνο αφορά θέματα διαφάνειας. Γιατί είναι μέλημα των πολιτών και επειδή είναι μέλημα των πολιτών, φυσικά ενδιαφέρει τον διαμεσολαβητή. Αναφέρθηκε ήδη η σημασία του νομοθέτη και της νομοθεσίας. Εμείς είμαστε παρατηρητές αυτής της νομοθεσίας. Ελπίζουμε ότι η νομοθετική αναθεώρηση πάντα θα μας οδηγήσει σε καλύτερη κατάσταση από αυτή από την οποία ξεκινήσαμε. Και αν υπάρξει τροποποίηση των σημερινών κανόνων, ελπίζουμε να είναι θετική η εξέλιξη και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ο Ομπούτσμαν πρέπει να σεβαστεί όμως τους κανόνες και πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα θεσμικά όργανα ε, ερμηνεύουν τους κανόνες με τον πιο διαφανή τρόπο που είναι δυνατόν στα πλαίσια των ορίων των κανόνων και να δούμε πέρα από τα αυστηρά όρια των, της νομοθεσίας για να δούμε αν τα θεσμικά όργανα μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Ε, ε, να είναι πιο φιλικά προς τον πολίτη για να, και να οικοδομήσουν αυτή την εμπιστοσύνη και θα σας δώσω και λίγα παραδείγματα για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ένα τελευταίο γενικό σχόλιο, ε, να επαναλάβω την παρατήρησα για, την, για το ρόλο του δικαστηρίου και τον ειδικό ρόλο του διαμεσολαβητή. Φυσικά ε, τα δικαστήρια εξετάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις που δεν μπορούν να εξετάσουν συστημικά θέματα. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό ένα δικαστήριο. Ο διαμεσολαβητής όμως δεν περιορίζεται από τέτοιου ε, περιορισμού. Μπορεί να δει τα συστημικά προβλήματα και να προτείνει συστημικέ λύσει αυτά. Και μπορεί να έχει ε, μια μακρο, μακρόπνοη θεώρηση και να καθοδηγήσει τα θεσμικά όργανα. Και αυτό είναι μια σημαντική προστιθέμενη αξία για το διαμεσολαβητή σε αυτό το πολύ σημαντικό τομέα. Μετά από αυτά τα γενικά σχόλια θα ήθελα να σταθώ σε ένα από τα δύο θέματα που ακούσαμε για το γενικό τεκμήριο που σημαίνει εάν ε, μία εξαίρεση ε, που προβλέπει η συνθήκη ισχύει. Αυτό δεν υπάρχει, δεν ανταναφέρει το ίδιο το δίκαιο, το, ο ίδιος ο νόμος. Το εντοπίζει το δικαστήριο. Ε, το Γενικό Τεκμήριο ότι υπάρχει μία ε, εξαίρεση, το αποφασίζει το δικαστήριο. Ε, Παραδείγματο χάρη, έχουμε ένα, μια, ένα κανονισμό που υιοθετήθηκε ε, και που λέει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα, ε, παραδείγματο χάρη στο δίκαιο ανταγωνισμού, θα πρέπει να παραμείνουν ε, μυστικά. Και έχετε από την άλλη τον 1049, έναν άλλον κανονισμό που βασίζεται σε ένα γενικό κανόνα ότι τα έγγραφα θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ε, επομένως, θα πρέπει να αντισταθμίσουμε τη θέληση του νομοθέτη που έχει εκφραστεί σε δύο διαφορετικά νομοθετικά κείμενα. Το πρόβλημα είναι και το έλεγαν και οι συναδελφοί μου και είναι πολύ σωστό αυτό, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και σωστά το θέσατε, ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα γενικά τεκμήρια ε, κινούνται και προς άλλους τομείς όπου δεν υπάρχει ε, τέτοια αντικρουόμενη νομοθεσία. Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επί παραβάση ή φερρυπίν σε σχέση με έγγραφα που ετοιμάζει η Κομισιόν και που οδηγούν σε προτάσεις ε, για νομοθεσία. Αυτή η επέκταση των γενικών τεκμηρίων ε, είναι, δημιουργεί ανησυχίε. Και γιατί το λέω αυτό. Για να σε ενημερώσω ότι ο διαμεσολαβητής δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα. Και αν ο διαμεσολαβητής βρει ότι τα θεσμικά όργανα προσπαθούν να εφαρμόσουν τα γενικά τεκμήρια σε τομείς όπου δεν υπάρχει σαφής τεκμηρίωση, σαφής, σαφής λόγος για να τα εφαρμόσουν, τότε ο διαμεσολαβητής θα ζητήσει από τα θεσμικά όργανα αυτά να λογοδοτήσουν για αυτό το πράγμα. Τα τελευταία χρόνια, Φερρυπίν, ο διαμεσολαβητής ε, ήρθε σε επαφή με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε, κλινικές, ε, σε μελέτες ε, κλινικών δοκιμών που είναι πολύ σημαντικές για τους πολίτες γιατί ε, μιλάνε με πολλές λεπτομέρειες γιατί ένα φάρμακο ας πούμε είναι ε, ασφαλές και αποτελεσματικό για, για τους ανθρώπους, για μας, για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας. Ευτυχώς ε, οι περισσότεροι από εμά δεν χρειάζεται να πάρουμε τα περισσότερα φάρμακα. Αλλά είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε ότι αυτά τα φάρμακα είναι ασφαλή και να εμπιστευόμαστε και τη διαδικασία με την οποία καταλήγουμε σε αυτήν την απόφαση. Είναι σημαντική αυτή η εμπιστοσύνη να υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία. Αρχικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμό Φαρμάκων είπε ότι υπήρχε ένα γενικό τεκμήριο ότι αυτά τα έγγραφα και αυτά τα έγγραφα δεν θα έπρεπε λοιπόν να δημοσιοποιηθούν. Ε, άλλαξε όμως τη θέση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και τον ευχαριστούμε γι' αυτό μετά από παρέμβαση του διαμεσολαβητή. Αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω. Ε, ο διαμεσολαβητής προσπαθεί να ασχοληθεί με θέματα ε, υπέρ της διαφάνειας, να προωθήσει τη διαφάνεια, ούτω ώστε ε, να βασιστούμε στον νόμο βέβαια, και αυτό αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του διαμεσολαβητή για αυτό το θέμα, ε, την πρόσβαση δηλαδή στις εκθέσεις ε, κλινικών δοκιμών ε, του φαρμάκου Μύρα, που είναι ένα φάρμακο που αφορά ρευματοπάθειες. Είναι ένα φάρμακο που πουλάει πάρα πολύ, χρησιμοποιείται ευρέω και πολύ σημαντικό και ο διαμεσολαβητής είπε καταρχάς δεν υπάρχει τέτοιο γενικό τεκμήριο ότι εφαρμόζεται η εξαίρεση, αλλά υπάρχει μάλιστα γενικό τεκμήριο ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται από την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών. Αντίθετα, το, το Γενικό Τεκμήριο ε, συνηγορεί υπέρ της, του άλλου επιχειρήματο, του αντίθετου επιχειρήματο. Και θα πρέπει ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, λέει ο Δημοσιοδητή, να εξετάσει πάντα εάν ε, το γενικό τεκμήριο ότι η δημοσιοποίηση, ας πούμε, αυτή είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντο και αν αυτό το δημόσιο συμφέρον είναι πολύ πιο σημαντικό οποιοδήποτε εμπορικό συμφέρον μπορεί να υπάρχει για τη μη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί αν μπορούμε να δεχτούμε. Και είναι ένα επιχείρημα αυτό, έτσι. Άκουσα και ανησυχίε για τα γενικά τεκμήρια. Αλλά αν δεχτούμε ότι υπάρχει ένα γενικό τεκμήριο ότι εφαρμόζεται η εξαίρεση, τότε θα πρέπει να δεχτούμε ότι σε άλλε περιπτώσει για συγκεκριμένες κατηγορίες εγγράφων υπάρχει το γενικό τεκμήριο ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται από την δημοσίευση, από την αποκάλυψη. Και αυτό το είπε ο δημοσιολαβητής σε μία πρόσφατη υπόθεση, λοιπόν. Και μάλιστα το είπε με πολύ σαφή λόγια, ότι η δημόσια υγεία θα πρέπει πάντα να είναι το πρώτο μέλημα πιο πάνω από τα εμπορικά συμφέροντα. Περνάω τώρα σε ένα άλλο θέμα που προσπάθησε ο διαμεσολαβητής να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια, να βασιστεί στα όσα λέει ο καονισμός, αλλά να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια. Μιλάμε για τη διαφάνεια των εγγράφων που ετοιμάζει το Eurogroup. Το Eurogroup δεν είναι ένας ευρωπαϊκός φορέας ή ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στενός πώς ε, ο κανονισμός 1049 δεν ισχύει για το Eurogroup και τα έγγραφα που παράγει. Αλλά πέστε το αυτό στους πολίτες που περιμένουν. Ε, για, για τους πολίτες το Eurogroup είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτού του ίδιου, αυτού του τύπου οι νομικίστικες ε, αιτιολογίες και νομικίστικα επιχειρήματα που δεν πείθουν τους πολίτες και δεν οικοδομούν εμπιστοσύνη. Ο διαμεσολαβητής στα πλαίσια μιας συνεργασίας ήρθε σε επαφή λοιπόν με τον πρόεδρο του Eurogroup και τον κύριο Ντάισεμπλουμ δηλαδή, και με χαρά λέμε ότι ε, είδαμε μια θετική απόκριση του Προέδρου του Eurogroup, του κύριου Ντάισεμπλουμ. Ε, είπε και αυτός με έμφαση ότι θα πρέπει να βοηθήσουν και αυτοί στην οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουν τη διαφάνεια. Δηλαδή, ε, μετά από την κίνηση του διαμεσολαβητή, δέχτηκε ότι πρέπει να βοηθήσουν τη διαφάνεια. Βέβαια, είπε το νομικίστικο επιχείρημα ότι υπάρχει ένα τεκμήριο, ας πούμε, που συνηγορεί υπέρ της μη αποκάλυψης. Εν πάση αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει ο διαμεσολαβητή. Δεν μπορεί να το κάνει όμω το δικαστήριο. Δεν μπορεί ένα δικαστήριο να κοιτάξει τέτοια θέματα από τη νομική σκοπιά. Αλλά το, ο διαμεσολαβητής φυσικά ε, έχει την εντολή να εξασφαλίζει την ε, εφαρμογή των κανόνων και το κάνουμε πάντα με μεγάλο ζήλο. Αλλά προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε και τη διαφάνεια. Να, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα τώρα που σχετίζεται με την ανησυχία της ε, Ευρωβουλευτού της κυρίας Εύη. Δεν θα μπω σε πολλέ λεπτομέρειε γιατί μίλησαν και οι συναδελφοί μου γι' αυτό. Θα ήθελα να σα πω όμω ποιο είναι ο ρόλο του διαμεσολαβητή στο θέμα αυτό. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι και εμεί είπαμε ότι σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές πληροφορίε, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα γενικό τεκμήριο σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ε, του δημοσίου συμφέροντος και κατά πόσο εξυπηρετείται από την ε, δημοσίευση των πληροφοριών. Προηγουμένως μίλησα για την πρόσβαση σε πληροφορίες ε, εκθέσεων που περιέχουν εκθέσεις για κλινικές δοκιμές. Το δικαστήριο μάλιστα ε, κινείται και προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, εξέφρασε και ε, συντένταξε και γνωμοδοτήσει προς την ε, κατεύθυνση αυτή. Ο διαμεσολαβητής το έχει κάνει εδώ και χρόνια. Ε, το πρόβλημα για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι ότι μερικές φορές κρατείται σε επίπεδο κρατών μελών και μερικές φορές κρατείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά ότι προφανώς ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής δουλεύει με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ε, και καλύπτει μόνο τα έγγραφα τα οποία ε, έχουν στη διάθεσή τους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπηρεσίες και οργανισμοί. Πάντως, υπάρχουν πολλά σημαντικά έγγραφα που σε αυτό επίπεδο, επίπεδο και εμπίπτουν ας στην εντολή του Διαμεσολαβητή και του Δικαστηρίου. Παραδείγματο χάρη, ο διαμεσολαβητή ασχολήθηκε με θέματα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που χρηματοδοτεί συχνά μεγάλα έργα υποδομή και που στα πλαίσια τη δουλειά τη ε, έχει έγγραφα που έλαβε από τα κράτη-μέλη για αυτά τα έργα, τα μεγάλα αυτά έργα υποδομών. Ε, εμείς ασχοληθήκαμε με υποθέσεις ε, εργοστασίων ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα στην Πολωνία. Ε, μετά την παρέμβαση του διαμεσολαβητή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είχε στη διάθεσή τη τέτοια έγγραφα, δέχτηκε να τα δημοσιοποιήσει. Είναι άλλο, υπάρχει ένα άλλο ε, περίπλοκο θέμα. Ε, κατά πόσον η Κομισιόν ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που έχει για διαδικασία παραβάση εναντίον κρατών μελών που δεν αποκαλύπτουν περιβαλλοντικές πληροφορίε που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό που είπαμε, αν δεν έχουμε επαρκή διαφάνεια σε επίπεδο κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ε, περιβαλλοντική ενημέρωση και περιβαλλοντικά στοιχεία, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανόνες σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν γίνεται. Άρα το θέμα τελικά ε, καταλήγει στο αν τα κράτη-μέλη συμμορφώνται με τις πληροφορίες, με τις υποχρεώσεις τους ό,τι αφορά την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαμεσολαβητής για το περιβάλλον είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με την Κομισιόν επίσης ε, για την ε, δημοσιοποίηση πληροφοριών σε ό,τι αφορά από θέματα τόνου που ψαρεύονται στη Μάλτα. Η Κομισιόν έχει σημαντικότατες εξουσίες ό,τι αφορά την, το περιβάλλον και τέτοια θέματα. Αυτές είναι οι, αυτή είναι η τομή όπου τα θεσμικά αυτά όργανα έχουν σημαντικό ρόλο και έχουν σημαντικές προφορίες για το περιβάλλον. Και εκεί ακριβώς ο διαμεσολαβητής κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε οι κανόνες οι συγκεκριμένοι να εφαρμόζονται σωστά. Μετά από αυτό που είπα προηγουμένως, για το Eurogroup θέλω να σας πω ότι ο διαμεσολαβητής ε, ήρθε σε επαφή με το Συμβούλιο για έγγραφα για την αξιολόγηση υποψηφίων ε, προκειμένου να αναλάβουν το αξίωμα του δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, στο ας πούμε, στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε τεράστιες συζητήσεις για τον διορισμό αυτών των ανθρώπων. Εμείς ούτε στο δαχτυλάκι των Αμερικανών δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, υπάρχουν αυτά τα έγγραφα που μιλούν για την αξιολόγηση των υποψηφίων και το σημαντικό ε, που πέτυχε η διαμεσολαβήτρια είναι να συμφωνήσει το Συμβούλιο ότι οι κανόνες για διαφάνεια ισχύουν σε αυτά τα, για αυτά τα έγγραφα. Το πρώτο τμήμα του επιχειρήματο ό,τι αφορά την πρόσβαση στην τεκμηρίωση είναι η συμφωνία ότι εφαρμόζονται, ότι ισχύουν αυτοί οι κανόνες. και ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Το δέχτηκε το Συμβούλιο. Στην αρχή ε, είχε ε, αμφιβολίες, αλλά τώρα συμφώνησε και δέχτηκε ότι το κοινό έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Θέλω να, ε, και επειδή θέλω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων και του κοινού, θα τελειώσω με το κάτωθι. Η πρόσβαση σε τεκμηρίωση που αφορά την νομοθετική διαδικασία. Ο κανονισμός, όταν μιλάει για αυτά τα έγγραφα, έχει ένα ευρύτατο ορισμό. Οποιαδήποτε έγγραφα που συνδέονται με την διαδικασία μέσω της οποίας ε, υιοθετούνται οι δεσμευτικοί κανόνες για τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει και διεθνείς συμφωνίες τεχνικός πώς, γιατί οι διεθνείς συμφωνίες είναι θαυμάσιο παράδειγμα και γιατί οδηγούν σε κανόνες που δεν διαφέρουν σε τίποτα σε ό,τι αφορά την ε, επίπτωσή τους ε, στα κράτη-μέλη και στους πολίτες, όπως, η νομοθεσία, ε, όπως και η νομοθεσία. Είναι ακριβώς το ίδιο. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό οι αρχές που αναφέρει ο κανονισμός, που λέει ότι ένα μεγαλύτερο επίπεδο διαφάνειας απαιτείται σε ό,τι αφορά αυτά τα έγγραφα, θα πρέπει να καλύπτει και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις που οδηγούν σε τέτοιου είδου αποτελέσματα. το χάρη το TTIP. Να γιατί είναι τόσο σημαντικό. Γιατί δεν διαφέρουν σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα από την συνήθη νομοθεσία. Και τα έγγραφα προκύπτουν από τη συνήθη νομοθεσία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, πρώτο πολύ σημαντικό που θέλω να πω. Και το δεύτερο, θέλω να το πω για τους ε, τριμερείς διαλόγους. Ε, συνεχίζονται τριμερείς διάλογοι ε, για το TTIP και και είμαστε χαρούμενοι που η Κομισιόν και άλλα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι ένα μεγαλύτερο επίπεδο διαφάνειας απαιτείται στη διαπραγματεύση στη ΤΥΠ. Ήδη άλλαξε νοοτροπία σε αυτήν την κατεύθυνση. Πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να δημοσιοποιηθούν τέτοια έγγραφα. Τώρα έχουμε πολύ μεγάλη αποκάλυψη εγγράφων και με συστημικό και δραστήριο, έτσι και ενεργό τρόπο. Ο κανονισμός 1049 αρχικά, αρχικά έτσι αναφέρεται με το θέμα ε, πρόσβαση στα έγγραφα κατόπιν ε, που γίνεται και γιατί ε, ενδεχομένως υπάρχει άρνηση. Το, το βασικό είναι όμως να υπάρχει έτσι αποκάλυψη υποφοριών ε, χωρίς να το ζητήσει κανένας. Να το κάνει το θεσμικό όργανο, α πούμε, από μόνο του. Ε, γιατί θα πρέπει να τα ζητήσει το κοινό. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν εκ Φυσικά δεν ε, απαγορεύεται κάποιος να ζητήσει ε, και επιπλέον έγραφα αν μια πολιτική έτσι υπέρ της ε, δημοσιοποίησης δεν είναι επαρκής, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει ως ιδιοφετηρία σε αυτή η πολιτική. Χαιρόμαστε λοιπόν για το αποτέλεσμα για το TTIP, χαιρόμαστε για τα αποτελέσματα για τους τριμμένους διαλόγους. Εμείς δεν έχουμε πάρει θέση ακόμα για αυτό το θέμα, ε, αλλά με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι το ε, ο διαμεσολαβητής χαίρεται που έχει καλή επαφή έτσι, με τα θεσμικά όργανα. Λάβαμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Ε, και εμείς έχουμε και δια, διαπραγματεύσεις επαφές με ε, άλλους φορείς παραδείγματος χάρη με την Γαλλική Βουλή, με το Γαλλικό Κοινοβούλιο, με, την, με τη Βρετανική Βουλή, με την Ολλανδική Βουλή. Γιατί βλέπουμε ότι και κρατικοί φορείς αναγνωρίζουν τη σημασία ε, διαφάνειας ε, γιατί η οικοδομή εμπιστοσύνη. Δεν θα πω τίποτα άλλο για τους τρομές διαλόγους γιατί το θέμα είναι εξελίξει. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω τις απόψεις του διαμεσολαβητή, της Emily O'Reilly. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Ρίγαν. Τώρα θα ακούσουμε δύο εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για την πρόσβαση αυτή. Η κυρία Έλεν Ντάμπισα πρώτη εκτελεστική διευθύντρια όσον αφορά το Accessing for Europe υπεύθυνη για την πλατφόρμα την διαδικτυακή όσον αφορά αυτό το έργο. Έχετε τον λόγο για 10 λεπτά παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Εντάξει αυτό το κουμπί. Πράγματι σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπή Αναφορών. Έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω κάποιες διαφάνειες Τρεις διαφάνειε έχω όλε όλε, αλλά θα ξεκινήσω. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή να παρίσταμε με ε, τους ανώτατους επικεφαλής ε, για αυτά τα θέματα σε αυτή τη συζήτηση. Στόχος μου είναι να συμπληρώσω κάποια από τα θέματα που προαναφέρθηκαν με πρακτικού χαρακτήρα παραδείγματα που θα δώσω. Μου ζητήθηκε να αναφέρω τι γίνεται με το Ask EU <clears throat> ε, όσον αφορά τα θέματα πρόσβασης με στόχο να είναι ευκολότερο για το κοινό να ζητήσουν, να απαιτήσουν διάθεση στοιχείων ενημέρωσης και πληροφόρησης. Αυτό σήμερα ακούσαμε για 3.000 αιτήματα όσον αφορά το Ask the EU. Και ένα από τα πράγματα που μάθαμε ποιο είναι. Πρώτα απ' όλα είναι θετικό το ότι είχαμε ενθαρρύνει τους ετούντες για να γνωρίζουν τα σχετικά και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ε, με βάση τη συνθήκη για να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπληρώνουμε την ιστοσελίδα μας με αυτό τον οδηγό για αυτές τις δυνατότητες. Είναι σημαντικό ότι οι απαντήσεις που δίνονται σε αιτήματα διατίθενται ευρύτερα, πράγμα το οποίο διασφαλίζει την διεύρυνση της διαφάνειας και επίσης ακολουθούμε τις διαδικασίες όσον αφορά τα αιτήματα υπό το πρίσμα της κοινωνίας των πολιτών. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για το πώς η πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα λειτουργεί στην πρακτική εφαρμογή. Δεν είναι τόσο απλό όσο ένα αίτημα και μια απάντηση αυτοματοποιημένα. Υπάρχει ένα ολόκληρο χρονικό πλαίσιο. Πολλές φορές προθεσμίες δεν είναι σεβαστές. Άλλες φορές υπάρχει εκ νέου αίτημα, παράταση, ως ένα χρονικό πλαίσιο. Έχουμε και αυτά τα μηνύματα όταν κάποιος πάει σε διακοπές που δεν απαντώνται. Και έχουμε εδώ ακριβώς το θέμα της άσκησης και δικαίωσης θεμελιώδους δικαιώματος. Μελετώντας τα θέματα αυτά μπορούμε να συντάξουμε συστάσεις, κάποιες από τις οποίες συνεισέφεραν σε αλλαγές ίσονος, ε, ελάσσονος σημασίας κάποια φορά, αλλά σημαντικό παρόλα αυτά θέμα. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αναγνώριση των ετοιμάτων από πλευράς του Συμβουλίου σε σχέση με τέτοιου είδους αιτήματα, βελτιώσεις. Μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε κάποια συστημικά προβλήματα που υφίστανται. Ένα από αυτά που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα καταχώρησης και καταγραφής. Είδαμε ότι πολλές φορές πρακτικά συνεδριάσεων είναι ανύπαρκτα. Και αυτό είναι μια πρόκληση, μεγάλη πρόκληση για τους κοσμήτορες. Μπορεί κανείς να ζητήσει έγγραφα, αλλά δεν μπορεί να ζητήσει γενικόλογα πληροφορίες. Αν μπορεί κανείς να φανταστεί τι συνέβη κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας λήψης απόφασης, δεν μπορεί απλώς να ζητήσει ένα, μια παρήθμιση συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα, διότι είναι απίθανο να υπάρχει κάποιος τέτοιος κατάλογος. Πώς γνωρίζει λοιπόν κανείς πότε έγιναν τέτοιες συνεδριάσεις, ώστε να προσπαθήσει να έχει πρόσβαση σε τέτοια έγγραφα τέτοιων συνεδριάσεων ή να έχει τα πρακτικά, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τέτοια πρακτικά δεν υφίστανται έχουμε και θέμα νομικών συμβουλών που προφορικά δινόντουσαν, πράγμα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Βλέπουμε ότι αποκλειστικός εμπιστευτικός χαρακτήρας εκ των ενόντων ad hoc εφαρμόζεται σε σχέση για παράδειγμα λέει με προκλήσεις όσον αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα και όσον αφορά υπαλλήλου ε, ε, που πρέπει να ε, μην αποκαλύπτουν στοιχεία. Και για παράδειγμα όταν έχουμε συνεδριάσεις π.χ. του Συμβουλίου σε, κάποια, σε κάποιες από τις ομάδες εργασίας κάποιοι υπάλληλοι κάποιων κρατών μελών ζήτησαν τα ονόματά τους να μην γνωστοποιηθούν ενώ άλλων στελεχών γνωστοποιήθηκαν βλέπουμε ένα παράλογο τρόπο. Εκείνοι που συμμετέχουν σε κάποια συνεδρίαση έχουν με κενό το όνομα του εκπροσώπου από την Λετωνία για παράδειγμα. Για ποιο λόγο να μην γνωστοποιείτε το όνομα ή τα στοιχεία ενός ε, στελέχους, ενός υπαλλήλου. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να είναι σαφές και κατανόητο. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να δει κανεί ποιο ποσοστό, σε ποιο ποσοστό συχνότητα ε, στον χρόνο συμβαίνουν τέτοια πράγματα, όμως παρόλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα για τα θέματα αυτά τα οποία είναι πρακτικού χαρακτήρα να πάρει κανείς, να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες βλέπουμε τι συμβαίνει. Άλλο αρνητικό, μια στιγμή, επόμενη διαφάνεια, μάλιστα επόμενη διαφάνεια είναι το δώρο της 9ης Μαΐου σε σχέση <coughs> με την άφηξη ε, αυτού του ε, μηνύματος, αυτού του δέματος ε, όσον αφορά τη βάση δεδομένων με τη, στην οποία καταχωρούνται στοιχεία. Θα ήθελα, θα επανέλθω σε αυτό να αναφέρω ότι εδώ υπάρχει, υπάρχουν αντιστάσεις και αρνητικές επιπτώσεις σε θέματα που προανέφεραν προλαλήσαντες, αντίσταση για να υπάρξει διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει και επιμένει η ταχυδρομική διεύθυνση κάθε ετούντος για διάθεση, για προσπάθεια πρόσβαση σε έγγραφα να καταχωρείται και να είναι δεδομένη. Δύο λόγοι εδώ, δύο λόγους επικαλούνται. Να γνωρίζουν λέει ότι οι ετούντες είναι αυθεντικά ετούντες ως άτομα, παρότι υπάρχει δυσκολία επαλήθευσης αν κάτι τέτοιο συμβαίνει ή όχι. Και διασφάλιση νομικής βεβαιότητας στην διάθεση πληροφοριών ηλεκτρονικά με email διατίθενται αυτές οι πληροφορίες. Μετά, μια εβδομάδα ή δέκα μέρες μετά, ή με τέτοιο πακέτο από το DHL, φτάνει η πληροφόρηση στο αντίστοιχο γραφείο ή στον ετούντα, στον πολίτη, στην οργάνωση, σύλλογο, δημοσιογράφο, οποιονδήποτε. Υπό το δικό μας πρίσμα αυτό αυξάνει όχι μόνο την αβεβαιότητα, αλλά δημιουργεί και δυσκολία όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο για την καταγραφή καταχώρηση ενός αιτήματο. Θα ξεκινάει αυτό από την ημερομηνία ενός ηλεκτρονικού μηνύματος ή αργότερα μεταγενέστερα με την άφηξη ενός δέματος ή πακέτου. Αυτό όντας δεδομένο, μία από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε βλέποντας το θέμα και τους κανονισμούς πρόσβασης ε, στοιχεία είναι πώς θα το λύσουμε. Χρειαζόμαστε λύσεις ε, του 21ου αιώνα για την επικοινωνία μεταξύ πολίτη και υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφάνεια είναι αυτή η διασύνδεση ακριβώς με τους πολίτες. Όταν περιπλέκονται όμως σε τέτοιο βαθμό αυτά τα πράγματα διοικητικά, αν θα πρέπει να είναι διαδικτυακά με email ή πώς και μετά μπορούν λέει, να σας απαντούν με το ταχυδρομείο, ε, πρέπει πολύ σοβαρά να ρωτήσουμε και να προβληματιστούμε πώς είναι δυνατόν να διευκολύνουμε το κοινό τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες όσον αφορά τα 500 τόσα εκατομμύρια πολίτες που μπορεί να έχουν τέτοια αιτήματα και απαιτήσει. Τώρα θα κάνω ένα άλμα περνώντας σε κάποιες από τις ενεξελίξει πρακτικές και περιπτώσεις που και αυτές καταδεικνύουν το πρόβλημα πως έχει. Στην πλατφόρμα μας ως EU ε, βλέπουμε ότι 60 ή 70% των ετοιμάτων την χάνουν απάντησης. Κατά το μάλλον ή των ικανοποιητικών απαντήσεων. Και βλέπουμε εδώ σε σχέση με το ποσοστό επιτυχίας εντός εισαγωγικών πολλές πληροφορίες διατίθενται. Εντάξει, όμως Βλέπουμε σημαντικές προκλήσεις ότι υφίστανται αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε εντό εισαγωγικών ευαίσθητα θέματα, sensitive issues. Και σε σχέση για παράδειγμα με το διορισμό δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο 10, καθορίσαμε τώρα ότι έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τέτοιες πληροφορίες Επόμενο βήμα. Ζητήσαμε την πληροφορία αυτή, δεν μας τη διέθεσαν. Τι πρέπει τώρα να γίνει, πώς θα διασφαλίσουμε συνέχεια. Τι τύπα, τις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων με τη ΣΥΠΑ. Τι γίνεται με την TTIP. Πού βρίσκεται η απόφαση σε σχέση με το ποιες πληροφορίες θα διατίθενται ή όχι. Από πού εκπηγάζει και ξεκινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα 28 κράτη-μέλη, επιβάλλεται ίσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των έξω από αυτή, σε αυτή την περίπτωση από τις ΣΥΠΑ Ποια είναι η αμφίδρομη δράση μεταξύ των ε, διαφορών εμπλεκομένων όσον αφορά τη διασφάλιση διαφάνειας στα διαφορετικά διαστρώματα και ε, επίπεδα που έχουμε. Η διαφορά είναι το, η ανείχνευση του πώς λειτουργεί η τράπεζα δεδομένων καταγραφή σε σχέση με τους 28 ε, επιτρόπους, ε, καταγραφή στοιχείων, δαπάνες από πλευράς τους που καταχωρούνται. Και τι είδαμε. Αυτό που θεωρούσαμε ότι θα ήταν απλό και εύκολο να καταδειχθεί, πώς δηλαδή, σε ποιο βαθμό είναι διασφαλισμένη αυτή η διαφάνεια σε σχέση με τους επιτρόπους πόσα διατίθενται ως κονδύλια για διανυκτερεύσεις, για στέγαση, αρνήθηκαν να μας δώσουν αυτές τις πληροφορίες δεχόμενοι να δώσουν μόνο κάποια στοιχεία αναέτος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα όμως ε, έφεσης ε, ε, ή προσφυγής και κατά τους τελευταίους μήνες ε, έχουμε και τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς αποθηκεύονται αυτά τα στοιχεία και αν θα ήταν ίσως δυνατόν να έχουμε εξατομικευμένα τα στοιχεία αυτά για ε, διάφορα στελέχη ή άτομα. Μας είπαν ότι δεν μπορούν να, να αντληθούν, να ανασυρθούν από τις τράπεζες δεδομένων. Και θα παίρνει 83 λέει ολόκληρες μέρες ε, για κάποιον υπάλληλο για να αντλήσει, να ανασύρει αυτά τα στοιχεία από αυτές τις τράπεζες δεδομένων. Δυσανάλογο δηλαδή ως ε, ε, επίπεδο επένδυσης. Λοιπόν έχουμε πράγματι πρόβλημα εδώ με τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες. Αν ουσιώδεις βασικές πληροφορίες που διασφαλίζουν την λογοδοσία για την δαπάνη δημοσίων κονδυλίων πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε πολλά κράτη-μέλη, πόσα δαπανώνται από τους επιμέρους υπουργούς για το ένα ή άλλο θέμα, αν αυτά είναι τόσο δύσκολο να διαφοροποιηθούν και να διαχωριστούν από τράπεζες δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απελπιστική κατάσταση. Και βλέπουμε ότι ως μια συμβιβαστική προσωρινή λύση σε δύο εβδομάδες να υποβάλλονται αυτά τα στοιχεία χωρίς όμως να περιορίζονται τα δικαιώματά μας άσκησης κάποια προσφυγή ή έφεσης. Αυτό μας πήρε 7 μήνες για να το καταφέρουμε και βλέπουμε σε σχέση με περίοδο 2 εβδομάδων για τη διάθεση αυτών των στοιχείων. Είναι απελπιστική κατάσταση, τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Περνάω στην τελευταία πρόκληση στο πρόσφατο αυτό πλαίσιο. Πολλοί από εμά κατά το πρόσφατο διάστημα είδαμε αυτή την ε, επίμαχη αφίσα για τη ροή προσφύγων στην Ευρώπη που δημιουργεί αυτή την εκστρατεία για το δημοψήφισμα στην Μεγάλη Βρετανία ε, σε κάμποσες μέρες από σήμερα και βλέπουμε ότι όταν έχουμε συμφωνίες μεταξύ για παράδειγμα όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία του Μαρτίου και όταν βλέπουμε ότι το γραφείο μας για την πρόσβαση access και για τα θέματα νομιμότητας ή όχι αυτής της συμφωνίας, σκεφτήκαμε ότι χρήσιμο θα ήταν να ζητούσαμε νομικές συμβουλές για το αν κάτι τέτοιο είναι θεμητό ή όχι. Γνωρίζουμε από νομοσυμβούλους ότι πολλές φορές είναι δύσκολο το να έχει κανείς μια τέτοια πλήρη περιεκτική νομική συμβουλή. Και μας είπαν ότι δεν υπάρχει μια τέτοια ένα πλαίσιο νομικών συμβουλών γιατί δεν υπάρχει λέει τέτοια συμφωνία. Πόσοι αναγνωρίζουν από εμά και το γνωρίζουν ότι δεν υπήρχε λέει δεν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Κανένα έγγραφο εκτός από το δημοσίευμα το οποίο γνωστοποιήθηκε στον τύπο. Και από εκπομπές εγώ άκουσα χθε το βράδυ από το BBC για αυτή τη συμφωνία ΕΕ Τουρκίας αναλύσαμε τις τρεις <clears throat> ευρύτερες πώλησης εφημερίδες και ανέφεραν οι περισσότερες στα περισσότερα δημοσιεύματα ότι υπάρχει λέει μια τέτοια συμφωνία και όμως δεν υπάρχει έγγραφο τέτοιας συμφωνίας. Κάτι όμως συνέβη το Μάρτιο αφού έγινε λέει μια συμφωνία και λήφθη απόφαση διάθεσης κονδυλίων στην Τουρκία. Ζητήσαμε λοιπόν νομική συμβουλή για αυτή τη διαδικασία. Υπήρχαν προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας και πρόσφατα μας αρνήθηκαν νομοσυμβουλές σε σχέση με την Επιτροπή για την χρήση τριών μόνο εξαιρέσεων. Χρήση εξαίρεσης για τις διεθνείς συμβάσεις και σχέσεις, λήψης απόφασης και προστασία νομικών συμβουλών σε εξέλιξη, σε θέματα υποεξέλιξη ε, για την ε, έγκριση ή όχι τέτοιων διαδικασιών. Συνεργαζόμαστε με ε, δικηγόρους νομοσυμβούλους για να μπορέσουμε να προσβάλλουμε αυτού του είδους τις αποφάσεις. Το θέμα εδώ υπό το πρίσμα της διαφάνειας είναι όταν μιλάμε για θέματα εμπιστοσύνης, εμπιστοσύνης κλίματος και περιβάλλοντος εμπιστοσύνης για την TTIP και θα ολοκληρώσω σε μισό λεπτό υπό το πρίσμα των πολιτών της ΕΕ για αυτό το αμφιλεγόμενο επίμαχο θέμα των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται και των διαδικασιών σε ένα κλίμα όπου υπάρχει μεγάλη τεράστια παραπληροφόρηση που διαχέεται για το τι κάνει λέει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την απειλή που διαδραματίζουν, που δημιουργούν λέει οι πρόσφυγες σε σχέση με εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να φοβόμαστε την απειλή. Για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να μάθουν τι συνέβη και τι συμφωνήθηκε και πώς θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια και από ποιον και από ποιον προϋπολογισμό θα αντληθούν. Είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν αυτά τα στοιχεία και σε αυτή την περίπτωση σε σχέση με την αντιμετώπιση των προσφύγων και πώς ελήφθη αυτή η απόφαση όλα αυτά υπογραμμίζουν τον κατεπήγοντα χαρακτήρα με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αυξήσουμε και βελτιώσουμε τα επίπεδα διαφάνειας που έχουμε ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η συμμετοχή και η λογοδοσία που θέλουμε να επιβληθεί και να επιτευθεί η απουσία της οποίας πραγματικά είναι επιζήμια στο σύνολο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τάρπισερ. Και σε πιο συγκεκριμένο θέμα, την ε, διαφάνεια και παροχή πληροφοριών σε θέματα περιβαλλοντικά, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Αναής Μπερτιέ από την οργάνωση Client Earth, που είναι και αναφέρουσα επιτρο... Ε, αναφοράς που εξετάστηκε από την Επιτροπή μας. Κυρία Μπερτιέ, έχετε 10 λεπτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και για την αναφορά μας. Ε, θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό που υπόθηκε πριν σχετικά με την ανάγκη για αναθεώρηση του ε, κανονισμού 1049. Θα το κάνω αυτό όμως ε, στην παρουσίασή μου. Συμφωνώ με την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, καθώς και την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νομολογίας. Ο 1049 είναι παλαιός πια αλλά Πιστεύουμε ότι ένα αίτημα σχετικά με το 1049 δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα στα θεσμικά όργανα σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι η αναθεώρηση θα κάνει αρκετή ζημιά. Θα επανέλθω όμως στο θέμα αυτό. υποβάλαμε αναφορά στην Επιτροπή σας ε, το 2012, η οποία ασχολείται με κάποιες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ε, της Κομισιόν με τον κανονισμό 1049, αλλά και με τις ε, διατάξεις για παροχή πληροφοριών της Σύμβασης του Όρχους. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσά, οι διατάξεις ε, της ε, σύμβασης έχουν εφαρμοστεί με τον κανονισμό του, Αρχούσε τον κανονισμό 1367 του 2006, που εφαρμόζει τη σύμβαση στα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς ε, και τους άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται πολύ σωστά και πολύ καλά ε, υπάρχει πολύ καλός ε, ορισμός ε, των περιβαλλοντικών θεμάτων και η σύμβαση του Όρχους, μάλλον ο κανονισμός του Όρχους εφαρμόζει πολύ σωστά αυτόν τον ορισμό και προχωράει ακόμα πιο πέρα όσον αφορά τις, τα ραδιενεργά απόβλητα. Ωστόσο, το πρόβλημα που έχουμε όσον αφορά την ε, ρύθμιση της ε, πληροφόρησης ε, από τον κανονισμό του όρχους. Το πρόβλημα είναι ότι όσον αφορά τις παρεκκλήσεις παραπέμπει στον κανονισμό 1049 που ισχύει για τις μη περιβαλλοντικές πληροφορίες. Έτσι λοιπόν δεν ρυθμίζεται σωστά η πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό του όρχους. Αυτό σημαίνει ότι όταν ζητάμε περιβαλλοντικές πληροφορίες, ισχύουν οι παρεκκλήσεις του κανονισμού 1049. Ποια ήταν λοιπόν τα προβλήματα που θίξαμε τότε και που πιστεύουμε ότι αποτελούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ε, με τον κανονισμό του Άρχους. Ε, σύμφωνα με τον κανονισμό 1049, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, είναι υποχρεωμένα να αρνηθούν πρόσβαση σε πληροφορίες εφόσον υπονομεύονται εμπορικά συμφέροντα. Σχετικό άρθρο επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να αρνηθούν την πρόσβαση σε πληροφορίες ε, εφόσον ε, θίγονται νόμιμα οικονομικά συμφέροντα ή εμπορικά συμφέροντα που προστατεύονται από τον νόμο. Οι παρεκκλήσεις ε, λοιπόν είναι πιο στενές στη μία περίπτωση από στην άλλη. Η προστασία των εμπορικών συμφερόντων, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας από τους λόγους που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το άρθρο 43... Επίσης ε, έχει γίνει η χρήση της παρέκκλησης, αλλά το άρθρο 43 έχει χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει την φήμη μιας εταιρείας. έχει χρησιμοποιηθεί, δηλαδή όχι επειδή οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικέ, αλλά για να μην ε, βλάψουν την ε, φήμη μιας εταιρεία. Αυτό δεν ε, μπορεί να γίνει αποδεκτό από εμά. Πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει το κοινό για να μπορεί να λαμβάνει εμπεριστατωμένες αποφάσεις, δεν θα πρέπει να προστατεύονται για να προστατευτεί η φήμη της εταιρείας. Επίσης, προβλέπεται στον 1049 ε η προστασία οικονομικών, ε, νομισματικών και οικονομικών πληροφοριών, κάτι που δεν αναφέρεται όμως στην σύμβαση του Όρχους. Μία μη κυβερνητική οργάνωση ήθελε πρόσβαση σε επιστολή που εστάλει από τον καγκελάριο της Γερμανίας τότε στη στον Επίτροπο Μεταφορών σχετικά με ε, βιότοπο και την ε, κατασκευή αεροδρομίου. Πρόκειται λοιπόν για περιβαλλοντική πληροφορία η οποία όμως δεν ε, δόθηκε επικαλούμενη αυτήν την παρέκκληση η οποία όμως δεν προβλέπεται στην σύμβαση του Όρχους. Δεν επιτρέπεται λοιπόν περιβαλλοντικές πληροφορίες να μην παρέχονται με αυτή τη βάση. Επίσης, ο 1049 προστατεύει τις έρευνες ποινικέ ή αστυνομικέ, αλλά η σύμβαση του όρχου όσον αφορά τι έρευνε προστατεύει μόνο ποινικέ και επιθαρχικέ περιπτώσει, όχι τι υπόλοιπε. Η συμβαση του ορχου οσον αφορα τις ερευνε προστατευει μονο ποινικε και επιθαρχικε περιπτωσεις οχι τις υπολοιπες η ευρωπαικη επιτροπη ομως δεν κάνει ποινικέ ή επιθαρχικές έρευνες. Ωστόσο, χρησιμοποιείται η παρέκκληση αυτή για να παρακρατηθούν όλε οι πληροφορίε που σχετίζονται με διαδικασίες επιπαραβάση, οι οποίε δεν είναι ούτε ποινικέ ούτε πειθαρχικέ. Και μάλιστα το δικαστήριο είπε σχετικά ότι η σύμβαση του άρχους δεν απευθύνεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Και επίσης η σύμβαση του άρχους δεν λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τι να σας πω, από νομικής πλευράς ε, το βρίσκω απολύτως αμφισβητήσιμο. Έχουμε το άρθρο 27 της Σύμβασης της Βιέννης που λέει ότι συμβαλόμενος σε διεθνή ε, σύμβαση δεν μπορεί να ε, επικαλείται ε, εθνικό νόμο για να μην τηρήσει τις διατάξεις της σύμβασης. Και ακριβώς αυτό γίνεται τώρα με τη σύμβαση του Όρχους. Είναι, δεσμικά, είναι νομικά δεσμευτική και για τα ευρωπαϊκά όργανα και για τα κράτη-μέλη. Επίσης, ο 1049 λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται πρόσβαση, πρέπει να αρνείται πρόσβαση. Είναι υποχρεωτική δηλαδή η διάταξη σε περιπτώσεις όπου η σύμβαση του Όρχου λέει ότι μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση. Θα θέλαμε πολύ λοιπόν ε, να εξετάσετε την ε, αναφορά μας. Επίσης, στήξαμε προβλήματα μη συμμόρφωσης με τον ε, κανονισμό 1049, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά δεν τηρεί τις προθεσμίες που προβλέπει ο κανονισμός 1049. Συστηματικά λοιπόν καθυστερεί πέρα από την προθεσμία που προβλέπεται στον 1049. Παραβιάζεται δηλαδή ο κανονισμός αυτός. Ε, ε, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ήδη έθιξε το θέμα, διότι ε, εμποδίζει την κοινωνία των πολιτών από το να έχει πληροφορίες εγκαίρως. Και αυτό αναφέρεται στην αναφορά μας όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν πριν. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το πλαίσιο της αναφοράς. Ο κανονισμός σε 1049 ε, συζητεί το τότε, καθώς και η αναδιατύπωσή του. Ε, λόγος να μην ζητήσουμε αναθεώρηση του κανονισμού είναι το ποια, ποιος ήταν ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχο είχε αποκλειστικά την αύξηση της εμπιστευτικότητας. Δεν υπήρχε καμία βελτίωση. υπό την Επιτροπή Παρόσο. Δεν, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί θα είναι καλύτερα τώρα υπό την Επιτροπή Γιούνκερ. Δεν έχουν... έχει βελτιωθεί η κατάσταση σήμερα. Αντιθέτως, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήταν να τροποποιηθεί ο ορισμός του εγγράφου. Ο ορισμός του εγγράφου είναι πολύ καλός, ε, διότι καλύπτει τα πάντα. Βάση δεδομένων, γραπτό ε, έγγραφο, όλα καλύπτονται από τον 1949. σε αντίθεση με τις διατάξεις της Σύμβασης του Όρχους, αλλά είναι καλός ορισμός αυτός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να περιορίσει τις κατηγορίες εγγράφων στις οποίες ε, θα έχει πρόσβαση ε, το κοινό. Θέλουν να επιβάλλουν περισσότερους περιορισμούς και τέλος ε, θέλαν να παρατείνουν τις χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να απαντάει σε αιτήματα. Όλα αυτά στόχο έχουν την αύξηση του καθεστώτος της και δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσε σήμερα να τους πείσει για το αντίθετο. Δεν έχω δει κανέναν αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να ε, υιοθετεί διαφορετική συμπεριφορά. Ε, γιατί κόλλησε η διαδικασία, ίσως ε, λόγω των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και επειδή υπήρχε εισηγητής ο, ο Μάικλ Κάσμαν, ο οποίος αγωνιζόταν για τη διαφάνεια και αμφισβητούσε κάθε λέξη της πρότασης. Αυτό δεν θα γινόταν απαραίτητα σήμερα. Εάν είχαμε εισηγητή του Κοινοβουλίου που να μην είναι υπέρ της ε, αυξημένης ε, διαφάνειας, μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και εν το Συμβούλιο προσπαθούσε να παρακάμψει την ε, νομολογία, όπως την υπόθεση Τούρκο. Ε, ζήτησε λοιπόν γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και αυτό αποτέλεσε σημαντικό βήμα οπισθοδρόμησης. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε πέντε αξιωματούχους που πίεζαν τους ε, εκπροσώπους ώστε το διοικητικό καθήκον να ορίζεται πολύ στενά, ώστε ο κανονισμός 1049 να μην καλύπτει πολλές ε, δραστηριότητες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αν συζητούσαμε σήμερα τον κανονισμό 1049 ότι θα έχει αλλάξει η κατάσταση. Νομίζω ότι μάλλον απλά ε, ε, έχει χειροτερέψει η κατάσταση. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα. Έχουμε το θεματολόγιο για την καλύτερη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχο έχει μια πιο διαφανή Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Σε αντίθεση με αυτό που ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να κάνει πιο διαφανή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ε, οι προσπάθειες αυτές καλύπτουν και την περιβαλλοντική νομοθεσία. Και επίσης, όπως υπόθηκε πριν, έχουμε τις μελέτες αντικτύπου, που είναι πολύ επίμαχο θέμα και που καθοδηγεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υιοθέτηση ή όχι ε, της νομοθεσίας. Και δυστυχώς ε, ισχύει τώρα το τεκμήριο της εμπιστευτικότητας από το δικαστήριο στις ε, μελέτες αντικτύπου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ε, πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά την ε, διαφάνεια. Οι συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών είναι εμπιστευτικές όπου συζητώνται οι τροπολογίες, οι τριμερείς διάλογοι όπου θέλουμε όχι μόνο να αυξήσει το Κοινοβούλιο την ε, διαφάνεια, αλλά και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει νόημα μόνο ο ένας από τους φορείς ε, να ε, αποκτήσει περισσότερη διαφάνεια. Έχει ζητηθεί η τριμερής διάλογη να είναι ανοιχτή προς το κοινό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δεν ε, ακολουθεί το δικό του ψήφισμα. Επίσης, όσον αφορά την ε, ΕΦΣΑ, την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, οι αποφάσεις σχετικά με το αν θα πρέπει να διτέθει στην αγορά ή όχι ένα συγκεκριμένο προϊόν διατροφής. Και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με εμπιστευτικό τρόπο κάτι που δεν συνάδει ούτε με την σύμβαση του Όρχους, ούτε με τον κανονισμό 1049. Είναι πολύ σημαντικό ανεξάρτητοι επιστήμονες ε, να εξηγούν τις ε, επιστημονικές ε, δοκιμές που έχουν γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει απλά σε ένα αναγνωστήριο να λάβει κανείς τις απαραίτητες πληροφορίες. Και ένας άλλος λόγος που επιμένουμε στην αναθεώρηση του 1049 όταν εξετάζει κανείς τέτοιες πολιτικές διαφάνειες. Ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πέρσι επανεξέτασε το ε, καθεστώς διαφάνειας της, ε, κάτι που έχουμε αμφισβητήσει και μάλιστα θα προσφύγουμε τώρα και στο δικαστήριο την υποθεσία αυτή. Έχουν συμπεριλάβει λοιπόν το ε, τεκμήριο τη εμπιστευτικότητα ότι αυτομάτω θεωρείται ε, ένα θέμα εμπιστευτικό εκτός ε, αν ισχύει το αντίθετο. Έτσι λοιπόν αυξάνεται η εμπιστευτικότητα και όχι η διαφάνεια. Άλλο στοιχείο είναι ότι πολύ πρόσφατα, τον Απρίλιο νομίζω, η οδηγία για τα για τις ε, εμπορικές ε, μυστικές πληροφορίες. Ε, η οδηγία αυτή ουσιαστικά ενθαρρύνει τις εταιρείε να θεωρούν εμπορικά απόρριτα ένα σωρό πληροφορίες και περιβαλλοντικές. Και υπάρχει περισσότερη ε, πληροφόρηση σχετικά με την σύμβαση του Όρχους, ε, όπου υπάρχει η διάταξη που λέει ότι δεν ε, μπορούν να καλύπτονται περιβαλλοντικές πληροφορίες, διότι κάτι τέτοιο είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Ε, επειδή υπήρχε αντίθεση από το Συμβούλιο, τελικά ε, έχουμε μόνο μια αιτιολογική σκέψη που αναφέρει την ε, σύμβαση του Όρχου. αλλά κάτι τέτοιο δεν αρκεί. Και η οδηγία αυτή δίνει περισσότερες δυνατότητες προσφυγής στο δικαστήριο για τις επιχειρήσεις. Και επειδή υπάρχει πίεση από μη κυβερνητικέ οργανώσει και δημοσιογράφου, οι επιχειρήσει θα το ξανασκέφτονται πρωτού δημοσιεύσουν πληροφορίε ε, εφόσον μπορούν να τις ε, παρουσιάσουν ως εμπορικό απόρριτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρνηθεί να ε, εκδώσει οδηγία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβαλλοντικά. Και οι σχετικές αποφάσεις θα βασίζονται αποκλειστικά στην ομολογία του δικαστηρίου και αυτή είναι η κατάσταση εντός ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι θέλουμε και πώς μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα. Όσον αφορά το μέλλον, λοιπόν, δεν υπάρχει ανάγκη να αναθεωρηθεί ο κανονισμός 1049, χρειάζεται να εφαρμόζεται καλύτερα. Και χρειάζεται καλύτερη νομική ερμηνεία του κανονισμού αυτού. Ωστόσο, μπορεί να αναθεωρηθεί ο κανονισμός του όρχους, κάτι που θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα, της, τα συμπεράσματα της Επιτροπής για τη συμμόρφωση με την ε, Σύμβαση του Όρχους. Πιστεύουμε πάντως ότι υπάρχει η νομική βάση να πιέσουμε ώστε να υπάρξει αναθεώρηση του κανονισμού του Όρχους, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη Σύμβαση του Όρχους. και επίσης ε, ώστε να ε, συμμορφώνονται οι διατάξεις σχετικά με την παροχή πληροφοριών ε, του κανονισμού με την σύμβαση. Σας ευχαριστώ και τώρα τελευταίος αγορητής θα, θα παρουσιάσει την Ολλανδική θέση της Ολλανδικής Προεδρίας την καλωσορίζουμε από πλευράς μόνιμης αντιπροσωπείας της Ολλανδίας για την δράση υπό την Ολλανδική Προεδρία υπέρ της διαφάνειας και της ελευθερίας πληροφόρησης. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά να παρίσταμε σήμερα, να μπορώ να πω δύο λόγια για το έργο της Ολλανδικής Προεδρίας για την προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας στην λήψη αποφάσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πολύ κοντά στις επιθυμίες μας, ε, στη δράση μας αυτό το θέμα για μας, όπως και για τους προλαλήσαντες η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενίσχυση της δημοκρατικής ε, νομιμότητας και θεμητότητας ε, απαιτεί αυτό το στοιχείο. Η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη βαίνουν εκ παραλλήλου. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει την υποστήριξη των πολιτών και πρέπει να είναι ανοιχτή και με διαφάνεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ολλανδική Προεδρία ήθελε και θέλει και μέχρι τέλους της Προεδρίας της ακόμα να βοηθήσει να καταστεί πιο διαφανή η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αυξηθεί η υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή νομιμότητα αλλά βήμα προς βήμα όλα αυτά, όλα αυτά. Πρέπει μια σταδιακή κλιμακούμενη πορεία βήμα προς βήμα να ακολουθηθεί για τη διασφάλεια της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Δεν θέλαμε επανάσταση στην διαφάνεια. Θέλαμε πραγματιστική, ρεαλιστική προσέγγιση, υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων πάντα σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ωστόσο, πρωτού υπησέθω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά αυτή τη βήμα προς βήμα προσέγγιση για τη διαφάνεια τη Ολλανδική Προεδρίας, δύο λόγια για τα θέματα διαφάνειας. Να υπογραμμίσω ότι για μας η διαφάνεια δεν είναι μόνο θέμα πρόσβαση σε έγγραφα και έντυπα. Η διαφάνεια επίσης αφορά το θέμα πόσο εύκολο είναι ή δεν είναι να βρει κανείς τις πληροφορίες και αν μπορεί κανείς εύληπτα να κατανοήσει τις πληροφορίες που διατίθενται. Η διαφάνεια είναι θέμα ιχνηλασιμότητας λοιπόν, ανείχνευσης μέχρι την πρόσβαση των πληροφοριών στα συναφή πλαίσια. Σήμερα είναι περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες από ό,τι οποτεδήποτε κατά το παρελθόν. Υπερβολικά πολλές πληροφορίες και δεν υπάρχει επαρκής χρόνος στη διάθεσή μας. Με τόσες πληροφορίες γύρω μας έχει κέρια σημασία να διοργανώσουμε το πλαίσιο εύληπτου τρόπου κατανόησης και άντλησης των πληροφοριών η Ευρώπη μπορεί να κερδίσει από την διάθεση, διοργάνωση και επεξήγηση αυτών των πληροφοριών. Οι λήψει αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνονται σε ένα ανοιχτό πλαίσιο, αλλά δεν το βλέπουν έτσι οι πολίτες και θεωρούν ότι υπάρχουν και στεγανά. Και παρότι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Δεν είναι αυτό ακριβώς το θέμα. Είναι το πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει σκληρά να εργαστούμε ώστε να γίνει πιο διαφανής η Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι οι πληροφορίες ε, πιο προσπελάσιμες. Ε, σε πιο ελεύθερη διάθεση. Πρέπει όμως εδώ να, γνωρίζουμε και τα όρια της διαφάνειας. Όπως σε όλες τις διαπραγματεύσεις, έτσι και στη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απαιτείται ένας βαθμός εμπιστευτικότητας. Για να διασφαλιστεί η περαιτέρω πορεία των διαπραγματεύσεων, επιτρέψτε μου μια σύγκριση. Ένας επικεφαλής, ε, για παράδειγμα, ε, μιας ομάδας σε σχέση με τα στοιχεία που έχει, Πολλά από αυτά θέλει να τα κρατήσει εμπιστευτικά για να είναι πιο αποτελεσματική επίδοση της ομάδας του. Όπως είπα στην αρχή, επικεντρωνόμαστε ως Ολλανδική Προεδρία σε πρακτικού χαρακτήρα βήματα και διαβήματα και όπου είναι δυνατόν πάντα σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, άλλες φορές με τα θεσμικά όργανα. Μικρά βήματα, βηματάκια παιδικά πολλές φορές, baby steps, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το στόχο είναι σημαντικό να γίνεται αυτό και από πλευρά των κρατών μελών. Για παράδειγμα, η προσοχή που δίνεται στη διαφάνεια όσον αφορά τη διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθετική αποδοτικότητα. Αυτό δείχνει την δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιωθούν τα θέματα διαφάνεια. Διαφορετικέ ε, απόψει και μελήματα, ανησυχίε υπάρχουν στα κράτη-μέλη για το ποια μορφή πρέπει να πάρουν όλα αυτά. Τα όρια, μέχρι πού θα φτάσουμε στη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με την δυναμική που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποστήριξη Πέρα από το ότι η διαφάνεια αποτελεί τμήμα των εργασιών μας, η Ολλανδία έχει συγκεκριμένες θέσεις για τη διαφάνεια και θεωρείται και προοδευτική και δεν είμαστε μόνοι μας εμείς σε αυτή τη θέση. Το 2015 συντάξαμε ένα non-paper, κοινό non-paper για τη διαφάνεια για την λήψη αποφάσεων με τη Δανία, Εστονία, Σλοβενία, Σουηδία και αυτό το έγγραφο αποτελεί τα θεμέλια αυτών που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας προωθούμε για αυτούς τους στόχους. Τώρα τέλος. Τι σημαίνει ακριβώς μια προσέγγιση βήμα προς βήμα. Πρώτα απ' όλα, να ασκεί κανείς αυτά τα οποία κηρύσσει, αυτά τα οποία λέει να τα τηρεί κανείς και να τα εφαρμόζει. Έτσι λοιπόν και για τις ε, δαπάνες ε, σχεδιαζόμενες και εκτελεστήσεις ε, θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα στοιχεία. Και από αναπληρωτού ε, εκπροσώπου και σε σχέση με την ε, τακτή βάση γνωστοποίησης ε, στοιχείων από πλευράς ε, της ε, αντιπροσώπευσης αυτό δείχνει μεγαλύτερη μέρημνα για την ικανοποίηση των μελημάτων των ομάδων που εμπλέκονται. Για πρώτη φορά είχαμε και μια εκδήλωση υιοθετώντα την προσέγγιση που από αποτελείται από δύο τμήματα. Την ε, ε, προσέγγιση ε, εύρους και την προσέγγιση εκδήλωσης. Έχουμε έτσι λοιπόν την εκδήλωση για να υπάρχει μεγαλύτερη γνωστοποίηση του πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αρκετές πρεσβείες της Ολλανδίας διοργάνωσαν αυτές τις εκδηλώσεις ε, Diplo Act, ε, διπλωματική δράση. Συνέρχονται διπλωμάτες ώστε να μπορέσουν ε, αυτές τις εκδηλώσεις να τις χρησιμοποιήσουν για την προαγωγή αυτών των στόχων. Μπόρεσαν λοιπόν στις 29 και 30 Απριλίου να συνέλθουν σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης ε, και μια διάσκεψη διοργανώθηκε κατά την 1η Ιουνίου. Τι σημαίνει μια unconference. Μόνο το θέμα ε, τέθηκε διαφάνεια. Η ημερήσια διάταξη αφέθηκε ελεύθερη στο να διαμορφωθεί από τους συμμετέχοντες με όλους τους εμπλεκόμενους ε, τους ε, αντιπροσώπους, αντιπροσωπείες, ε, συμβούλους για πολιτική, συμβούλους για θέματα πληροφορικής και τεχνολογιών. Όλοι είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν σε ένα ανοιχτό διάλογο για θέματα ευρωπαϊκής διαφάνειας. Επίσης προαναγγέλθηκε το έργο σε δράση μας που δείχνει ποιες δράσεις από το Συμβούλιο υπό συγκεκριμένη σύνθεση τηλέφωνο που παρισέφρισε συνεχίζει συμπεριλαμβάνοντας τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία δεν χρειάζεται τώρα να συμπεριληφθούν ε, πιο εξειδικεμένα. Όλα αυτά δείχνουν το δυναμικό αυτών των ανοιχτών ημερίδων τι μπορεί να γίνει ώστε να γίνουν πιο προσπελάσιμα και πιο φιλικά για τους χρήστες αυτά τα στοιχεία. Μια και μπορεί να θεωρηθεί γενικόλογο αυτό το πλαίσιο, έχουμε και ένα σύντομο βίντεο που θα ήθελα να σας παρουσιάσω και που μπορεί να ενημερώσει σχετικά. Για δείτε το.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 Για να συνεχίσω μετά από αυτή την παρουσίαση για την προσέγγιση βήμα προς βήμα. Συμπεριλαμβάνουμε τον χαρακτηρισμό εγγράφων στην ημερήσια διάταξη. με την Προεδρία μας, συνειδητοποίησαμε ότι δεν μπορούσαμε να πούμε ακριβώς πότε και γιατί έχουν χαρακτηριστεί κάποια ε, έγγραφα ε, περιορισμένης ε, ε, αποκάλυψης ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα, για τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για το λιμιτέ για τον περιορισμένο χαρακτήρα αυτών των εγγράφων. Υπό την Προεδρία μας στόχος μας ήταν να πάψει να ισχύει ο χαρακτηρισμός λιμιτέ για αυτά τα έγγραφα το δυνατόν ταχύτερα, όταν δηλαδή θα έχουν πλέον συζητηθεί στην Κορεπέρ, μετά να μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Και έτσι δημοσιοποιήθηκε πληροφόρηση που δείχνει περισσότερα στοιχεία για, αυτά, για αυτή την υπόθεση. Καταδεικνύεται ότι δύο τρίτα των στοιχείων των εγγράφων που είχαν χρησιμοποιηθεί διανέμονται πλέον, είναι διαθέσιμα ε, για το κοινό και επίσης σε σχέση με τις, ε, τα προκατακτικά, την προκατακτική φάση εργασιών όπου αποτελούν βάση για τις διαπραγματεύσεις ε, ή αντανακλούν την πρόοδο σε συγκεκριμένα θέματα αυτά θα πρέπει να παράγονται ως ε, έγγραφα σημαντικού χαρακτήρα και πρέπει να αναφέρονται και να καταγράφονται καταγεγραμμένα σε καταλόγους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να συνεισφέρουμε ενώ θα υπάρχει το θέμα της εμπιστευτικότητας να μπορούν παρόλα αυτά να γνωστοποιούνται στοιχεία σε σχέση με το 1049 και ένα τέτοιο αίτημα σε πρόσβαση για, ε, σε έγγραφα limite ε, εξετάζεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ε, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ευαισθησίας του φακέλου, το είδος ε, του εγγράφου και το ε, πώς θα μπορούσε να ελευθερωθεί ή όχι. 84% ενδεικτικά εγγράφων που σχετίζονται με ενεξελίξει νομοθετικές διαδικασίες που εκδόθηκαν το 2015 απελευθερώθηκαν μετά από αίτημά μας σε σχέση με το 1049. 84% δεν είναι κακή επίδοση καθόλου αυτή. Επίσης όσον αφορά την ημερήσια διάταξη της ομάδας εργασίας μετά από αίτημα της Ολλανδικής Προεδρίας υπήρξε το αίτημα να εξεταστεί η επίπτωση όσον αφορά την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τέτοιου είδους θέματα. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την δημόσια πρόσβαση σε τέτοιου είδους έγγραφα πρόσβαση σε έγγραφα των κρατών μελών και συνένεσε το Συμβούλιο να συνεχίσει η εξέταση αυτού του θέματος υπό τις υποεξέλιξη διαδικασίες νομικές παρότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση σε σχέση με κράτη-μέλη που επισημαίνουν την τοποθέτησή τους. Η αξιολόγηση έδειξε ότι αυτή η συμφωνία και τα όσα συνέβησαν μετά την ε, νομολογία του ε, δικαστηρίου δεν συνεισέφεραν σε μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τον τρόπο εργασίας από πλευρά του Συμβουλίου. Και ενώ δεν υπάρχουν προδιαγραφές ε, και γνώμονες, ε, δεν υπάρχει και σαφής ένδειξη ότι υπάρχει μείωση σε σχέση με την ε, περίπτωση αυτή. Εδώ πρέπει να αναφερθεί επίσης η αναδιατύπωση του κανονισμού 1049 που ήδη προαναφέρθηκε από προλαλήσαντες φαίνεται ότι υπάρχει πολύ περιορισμένο φάσμα να μπορέσει να προαθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο. Υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές απόψεων ε, μεταξύ των εμπλεκομένων που παρακολύουν αυτή την επικαιροποίηση ή ε, αλλαγή. Και έτσι λοιπόν αυτό δείχνει το τι εμπλέκει το 1049. Ωστόσο, από πλευράς των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει προσπάθεια να προχωρήσουμε. Εδώ θέλω να αναφέρω τις διαφορετικές προτάσεις υπό τον πρόεδρο της ε, Ευρωομάδας Eurogroup, κύριο Μπλουμ, για την προαγωγή της διαφάνειας. Όπως αποφασίστηκε τον Φεβρουάριο 2016, η ημερήσια διάταξη της Ευρωομάδας θα δημοσιοποιείται πριν από τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και μετά από τη συνεδρίαση θα μπορούν να γνωστοποιούνται συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω να ευχαριστήσω τη διαμεσολαβήτρια για την δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων. Δεν έχει καθοριστεί τελεσίδικα η ημερήσια διάταξη. Η διαφάνεια και πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση όλων των πτυχών διαφάνειας για την καλύτερη νομική, ε, νομοθετική εργασία θα πρέπει να μπορέσει να προωθεί Για να διευκολυνθεί η συζήτηση, η Ολλανδική Προεδρία συνέταξε ένα δημόσιο ε, σημείωμα σε σχέση με την προσέγγιση από το Συμβούλιο της χρήσης ε, κοινών τέτοιων δυνατοτήτων πρόσβασης ε, σε πληροφορίες με άμεσο γοργό τρόπο που θα προσαρμόζει σε σχέση με τις ανάγκες που υφίστανται περισσότερη διαφάνεια τριμερών διαλόγων σε σχέση και με την έκβαση των ίδιων των ε, τριμερών διαλόγων και σε σχέση με την ε, υλοποίηση των κατεκτέλεση πράξεων ε, και των ημερησίων διατάξεων. Φυσικά η υλοποίηση των διατάξεων για τη βελτιωμένη νομοθετική αποδοτικότητα είναι κάτι που θα παρακολουθήσουμε σε σχέση με θέματα διαφάνειας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα. Νομίζω έχω ξεπεράσει ήδη τα 10 λεπτά του χρόνου που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να σας έδωσα κάποια στοιχεία να κατανοήσετε την προσέγγιση της Ολλανδικής Προεδρίας κατά τους προηγούμενους 6 μήνες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Θα ήθελα μιλήσω πολωνικά. Με βοηθήσει η διερμηνία. Ευχαριστώ. Που... Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση τώρα. Ποιο θέλει να θέσει ερωτήσει να κάνει παρατηρήσεις. Κυρία Καμπεθόν. Ευχαριστώ. Έχω ξαναζητήσει το λόγο. Ε, θα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους, για αυτό το σημαντικό θέμα. Ε, είναι σημαντικό για να εμβαθύνουμε την δημοκρατία. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια που ζητάνε οι πολίτες και πολύ σωστά τη ζητάνε. Θα ήθελα να σταθώ σε μία από τις παρεμβάσεις που άκουσα και ένα συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό που είπε Ε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας ε, για τις, τις εκθέσεις από τις κλινικές δοκιμές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήθελα σε κάποια φάση να το πω και στην ίδια τη διαμεσολαβήτρια. Για το, το θέμα των φαρμάκων υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον που σημαίνει προστασία της υγείας. Ε, στην Ευρώπη έχουμε τα κράτη-μέλη που εξασφαλίζουν αυτό το δικαίωμα και από την άλλη ε, τα συμφέροντα μιας αγοράς, έτσι, που μπορεί να, το φάρμακο από μια σκοπιά μπορεί να θεωρηθεί ένα καταναλωτικό αγαθό, όπως τα άλλα. Ε, νομίζω ότι η σχέση αυτή είναι εντελώ ε, αδιαφανή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, ισορροπία ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και στο ιδιωτικό συμφέρον. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές ε, για να εξασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία. Πρέπει να είναι ανοιχτή η επιστήμη και θα θέλαμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την συζήτηση για το θέμα της, που είναι ιατρικό θέμα και συνεισφέροντας σε αυτό το ζήτημα των φαρμάκων. Ε, υπάρχει εδώ το θέμα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν ε, παράγεται ένα προϊόν, ε, τα μυστικά του προστατεύονται από το δίπλωμα βρεσιτεχνίας Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πολύ σημαντικά δεδομένα γύρω από τα φάρμακα. Για λόγους δημόσιας υγείας. Ε, πρέπει να δούμε τι ποιότητα έχουν αυτά τα φάρμακα. Είναι σημαντικό αυτό. Ε, επίσης είναι σημαντικό να δούμε πώς καθορίζονται οι τιμές κάποιων φαρμάκων, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και σε δικές μας χώρες λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είναι... Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχαμε διάφορα προβλήματα με διάφορα φάρμακα, ας πούμε τα φάρμακα κάτι υπατήτητα σε ε, που κατηγορούνται ε, ότι είναι καρκινογόνα. Επίσης, ο οργανισμός που δίνει τις άδειες για τα φάρμακα εμπλέκεται σε όλη αυτή τη συζήτηση. Ε, θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν συγκρούσεις ε, συμφερόντων. Δεν, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχουν. Ε, είναι σημαντικό επίσης να ερευνήσουμε το θέμα της χρηματοδότησης. Αν η χρηματοδότηση εξασφαλίζει αυτή την ασφάλεια και την ισορροπία ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο συμφέρον. Ο οργανισμός Φαρμάκο θα πρέπει να προάγει το δημόσιο συμφέρον και να εξασφαλίσει ότι δεν δημιουργούνται συγκρούσεις συμφερόντων λόγω της ε, ιδιωτικής ε, χρηματοδότησης. Ε, μερικές φορές η οι φαρμακοβιομηχανίες μέσω των φόρων που πληρώνουν εξαγοράζουν ε, ουσιαστικά τις άδειε που τους δίνονται. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Και είναι σημαντικό και ο διαμεσολαβητή να παίξει αυτό το ρόλο για να εξασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό συμφέρον. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Μερικές φορές με θλίψη ακούμε να υποστηρίζουν και άλλοι τις δικές σου, να ακούς να υποστηρίζουν και άλλοι τις δικές σου απόψεις. Ορισμένοι λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον 1049, τον κανονισμό 1049, αντί να τον επικαιροποιήσουμε. Πρέπει να βρούμε και να εξετάσουμε τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Αυτά τα λέω προς τον εκπρόσωπο της διαμεσολαβήτριας. Εγώ είμαι ο νησιώδης εισηγητής για την εφαρμογή α, της σύμβασης του Άρχους το 2006 και ήμουν και σκιώδης εισηγήτρια για τον κανονισμό που αφορούσε τη διαφάνεια των κλινικών δοκιμών. Βλέπουμε με θλίψη ότι το πεδίο εφαρμογή ε, περιορίζεται. Έχουμε την αίσθηση ότι κάνουμε βήματα προ τα πίσω ότι να προωθήσουμε κάποια συμφέροντα, διαφάνεια κλπ. Επίση, έχουμε την αίσθηση ότι το δικαστήριο δεν είναι αρκετά ισχυρό για να μα βοηθήσει. Δεν ξέρω τι νομικά εργαλεία έχουμε στα χέρια μα Τι εργαλεία μας δίνει η χάρτα ή η συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, νομίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μιλάει για το, τα πρωταρχικά α, δικαιώματα υγείας, α, περιβαλλοντικά κτλ. Έναντι των ε, εμπορικών συμφερόντων. Νομίζω ότι τα έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα επιχειρήματα και τα, τα εργαλεία που δίνει η ίδια η συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, ο διαμεσολαβητής στο παρελθόν. Νομίζω ότι ενώ κάναμε κάποια βήματα προς σωστή κατεύθυνση, τώρα κάνουμε βήματα από τα πίσω για τις τιμές ας πούμε των φαρμάκων. Πρέπει το Κοινοβούλιο να βοηθήσει. Πρέπει να καταλάβουμε τι εργαλεία έχουμε στα χέρια μας, ούτω ώστε να αναγκάσουμε την Κομισιόν να φτιάξει μια σωστή νομοθεσία που να σέβεται τη συνθήκη, που είναι το βασικό μας ε, νομικό εργαλείο, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Δεν θα πρέπει συνέχεια να οπισθοχωρούμε, να μειώνεται η διαφάνεια να αποθαρρύνονται οι πολίτες. Ο 1049 βάζει ε, κάποια όρια στην πληροφορία ε, και αυτό το έλεγε και η παλιά σύμβαση του Άρχους. Ήταν μια απόπειρα για να περιορίσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αντίθετα τώρα έχουμε και το, τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ισχύει η Χάρτα ε, και η Χάρτα είναι τμήμα του ενωσιακού δικαίου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ισχύει. Χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά. Γιατί οι δυνάμεις που είναι ενάντια στη διαφάνεια είναι πολύ ισχυρές. Θυμάμαι κάποιον από την Κομισιόν, ο οποίο ήξερε πάρα πολλά για την παλιά σύμβαση Άρχου. Και ενώ ήξερε πάρα πολλά και ήταν υπέρ της διαφάνειας, τον απομάκρυνα από τη Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο. Περιβάλλοντος. Αυτές οι ισχυρέ δυνάμεις είναι κοντόθωρες, μιοπικές και προασπίζουν τα εμπορικά συμφέροντα καθαρά. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων τώρα γίνεται όλο και πιο αδιαφανής. Ε, ταλανίζεται από συγκρούσεις συμφερόντων. Ε, και εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πρέπει να μας βοηθήσουν αυτοί που ξέρουν για να χρησιμοποιήσουμε τα νομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιπαλέψουμε αυτές τις ισχυρές σκοτεινές δυνάμεις που είναι ενάντια στη διαφάνεια. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Ε, νομίζω ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα με τη σειρά των ομιλητών. Σας ευχαριστώ για αυτού, τον προβληματισμό που μας παρουσιάζεται. Είμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση έχουμε αυτές τις α, ισχυρές ε, σκοτεινές δυνάμεις κατά της διαφάνειας. Από την άλλη βλέπω ότι στο Κοινοβούλιο ε, υπάρχουν πάρα πολλοί υποστηρικτέ και θειασότες της α, διαφάνειας σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Και συχνά ε, γίνονται εκδηλώσεις για την διαφάνεια, την ακαιρεότητα και τη λογοδοσία. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες της δημοκρατίας και το Κοινοβούλιο τους προωθεί. Νομίζω ότι είμαστε Πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί εμείς στο Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνω ότι οι προτάσει που έγιναν ε, είναι προς την κατεύθυνση του να φτιάξει ένα μοντέλο το Κοινοβούλιο ε, για να αναθεωρήσουμε τον 1049. Ε, με βάση την ομολογία και την νομική εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει, τα τελευταία 15 χρόνια, ακριβώς 15 χρόνια, από το 10, από τότε που φτιάξαμε τον 1049, τότε επί Σουηδικής Προεδρίας. Εγώ στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είμαι υπεύθυνη για την πρόθεση αυτής της πρότασης μιας ανοιχτής, ανεξάρτητης και αποτελεσματικής ε, ευρωπαϊκής υπαλληλίας. Ε, αναφέρεται και στο άρθρο ε, 2.98 της συνδίκης της Λισαβόνας, δεν έχει υπάρξει βέβαια δεύτερο γενναίες δίκαιο. Εμείς είχαμε συντάξει ε, ένα κανονισμό με ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες. Ο καθηγητής Κέρτιν είχε εμπλακεί, αν, δεν θυμάμαι, καλά τότε, ε, και βοηθήσαμε έτσι την Κομισιόν. Αλλά είναι, είναι και ώρα νομίζω να γίνουμε πολύ πιο επιθετικοί. Και χαίρομαι που η Ολλανδική Προεδρία μέσω του non-paper, το οποίο ελπίζω να είναι δημόσιο, ε, γιατί όταν το υιοθετήσατε τον Απρίλιο του 2015, ο, το υιοθετήσαν έξι χώρες, ονομαζόταν non-paper. Τουλάχιστον αυτές οι έξι χώρες θα πρέπει τώρα να συνεργαστούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθήσουμε την πραγματική και ουσιαστική και ρηξικέλευτη αναθεώρηση του 1049 ε, και να προωθήσουμε επίσης το δίκαιο για μια ανοιχτή, ε, αποτελεσματική, ανεξάρτητη ευρωπαϊκή διοίκηση. Τα ελλείμματα που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι τα εξή. Αυτά τα νομοθετικά κείμενα δημιουργούν τροχοπέδι και στο Κοινοβούλιο. Ακόμα και η κυρία Άουκεν, την οποία σέβομαι πάρα πολύ, ε, πιστεύει ε, ότι, ακόμα και εκείνη πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο κερδίζει από ένα κάποιο βαθμό μυστικότητας. Υπάρχουν διάφοροι ευρωβουλευτές όμως α, που πιστεύουν ότι το κοινοβούλιο δεν πρέπει να είναι 100% ανοιχτό στους διαλόγους ε, τους Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάρκεια ανάμεσα στα νομοθετικά κείμενα και στα υπόλοιπα κείμενα. Ε, υπάρχει ένα κενό εδώ για, στην εφαρμογή. Ε, Κοιτάξτε την έκθεση που υιοθετήθηκε το Κοινοβούλιο πριν από κάνα δύο μήνες για αυτά τα θέματα που εκφράζει βασικά, βασικές απόψεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα έγγραφα των τριμμένων διαλόγων. Και περιμένοντας την, το αποτέλεσμα της έρευνας του διαμεσολαβητή, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι τα έγγραφα των τριμμένων διαλόγων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα υπόλοιπα νομοθετικά κείμενα. Να σας πω και τη δική μου εμπειρία από τη στιγμή που τέσσερι ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων κοιμών ε, τίμασαν ένα έγγραφο για την πρόσβαση σε επιστημονική έρευνα, το βάλαμε και στην ιστοσελίδα, όπου η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Τροφίμων ε, βασίζονται για να αξιολογήσουν ε, διάφορα πιτοφάρμακα. Η τελική απόφαση θα ληφθεί αυτή την εβδομάδα από μια επιτροπή προσφυγών, γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν τεχνική επιτροπή. Αυτό που γίνεται είναι ότι η πρόεδρο, συμφωνώ με αυτό που είπε η πρόεδρο ε, Βίξτρομ, ε, για το θέμα τη εμπιστοσύνη. Ακόμα και ο επίτροπο αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στην κοινωνία και τι αρχέ, ε, οι οποίε δίνουν και τι άδειε για αυτέ τι ουσίε. Και έμεσα συμφώνησε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη πρόσβαση στα έγγραφα και στην τεκμηρίωση. Νομίζω ότι η εμπειρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων μπορεί να χρησιμεύσει εδώ. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα αιτήματα των πολιτών για πρόσβαση σε πληροφορίες. Εδώ υπάρχουν τρία ελλείμματα θα έλεγα. Η Κομισιόν καταρχάς, όπως αναφέρθηκε και από άλλους, είναι αυτός που έρχεται σε επαφή με τον Ετούντα προσπαθεί να τον καταλάβει καλύτερα, ε, αλλά νομίζω ότι η Κομισιόν και η ΕΦΣΑ μπερδεύονται ε, με αυτή την αρχή του δικαιώματος του δημιουργού. Για το αν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Η Κομισιόν μας είπε ότι είναι σε επαφή, μιλάει στους δημιουργούς ε, και στους ερευνητές, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν αποφασίζουν οι δημιουργοί. Αποφασίζει ένας φορέας. Και το δεύτερο είναι ότι κατά διάρκεια αυτή τη επαφή ε, και αλληλογραφία, και ενώ περιμέναμε την πρώτη απάντηση, προσφέρθηκε η Κομισιόν να μα να μας προσφέρει τη μέθοδο της ανάγνωσης μόνο. Όχι, όλο επεκτείνεται αυτή η μέθοδο. Στις αρχές με τον 1049 είχαμε αποφασίσει ε, ε, να αντιμετωπίσουμε... Εμάς δεν μας άρεσαν τώρα, τότε τα ε, εμπιστευτικά έγγραφα, αλλά προσπαθήσαμε να τα πιέσουμε μέσω αυτής της μεθόδου. Τώρα, βλέπουμε ότι τα έγγραφα του TTIP είναι ε, διαθέσιμα στους ευρωβουλευτές αλλά και στους εθνικούς βουλευτές μόνο σε ε, ειδικέ αίθουσε ανάγνωσης. Υπάρχει μόνο αυτή η μέθοδος της ανάγνωσης. Δεν πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει πραγματική πρόσβαση σε πολλά έγγραφα τα οποία ε, μπορούμε να τα διαβάσουμε απλώς σε συγκεκριμένους χώρους. Ε, που είναι το όριο τελικά, ειδικά σε διαπραγματεύσεις <coughs> ε, βασικά ε, μας υπαγορεύει η Αμερική τι θα κάνουμε. Η Επίτροπος Μάστομα έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά στην πραγματικότητα ε, απαρνήθηκε τη σημασία του καονισμου 1049 γιατί και συμφώνησε με τους Αμερικανούς ότι υπάρχει ένα όριστο τι μπορούν να πετύχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν είναι καθόλου κομψή η αντιμετώπιση των ετοιμάτων στα πλαίσια του 1049 από τις αρχές ε, και μην ξεχνάμε ότι το δίκαιο για την ανεξάρτητη ανοιχτή και διαφανή και αποτελεσματική ε, ευρωϊπαλληλία μπορεί να βοηθήσει. Θα πρέπει οι κανόνες αυτοί να ισχύουν για όλους τους ευρωπαϊκούς φορείς για τους, να ισχύουν για τους Ευρωπαίους πολίτες, για όλους τους ενδιαφερόμενους, ούτως ώστε οι πολίτες να καταλαβαίνουν καλύτερα ποια είναι η διαδικασία για να υποβάλουν έτοιμα α, πρόσβαση σε έγγραφα που κατέχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο κύριος Γιάννη. Μάλιστα, ευχαριστώ. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη. Λόγω άλλων ανελημμένων υποχρεώσεων ακροάσεων δεν μπόρεσα να παραστώ. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα μπορούσε κανείς να το να πει ότι από μακριά συμφωνούμε όλοι. Κανείς δεν έχει καμιά αντίρρηση για διαφάνεια. Μπορεί ίσως να παρηγορήσει να πω ότι σε σχέση με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων ζηλεύουμε καμιά φορά σε σχέση με το, μας ζηλεύουν σε σχέση με το επίπεδο διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την γερμανική ας το πω έτσι επίδοση συγκρίνοντας τα πράγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Αν αποσαφινιστούν αυτά, ίσως μπορέσουμε ταχύτερα να συμφωνήσουμε. Πρώτη ερώτηση. Υπάρχουν όρια διαφάνειας. Αν καθορίζαμε αυτά τα όρια, ίσως θα μπορούσαν τα θεσμικά όργανα γοργότερα να συμφωνήσουν σε σχέση με θέματα απορρίτου ή αποκάλυψης απορρίτου από πληροφοριοδότες δεν έχουμε κανένα κέρδος όταν οι πιο σημαντικές πληροφορίες παραμένουν εκτός εκτός πρόσβασης ε, των ε, οργάνων μας, των θεσμικών οργάνων. Ποιο είναι το κέρδος. Παράδειγμα, ένα παράδειγμα. Καμιά φορά πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ανταλλαγέ. Ε, αν δεν μπορούν να διεξαχθούν τέτοιες, τέτοιες ανταλλαγές, τότε δεν είναι δυνατόν να, ε, να πετύχουμε τίποτα, μια και τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται. Υπάρχουν όρια λοιπόν στη διαφάνεια. Να καθορίσουμε αυτά τα όρια πρώτα. Και δεύτερον, το θέμα του ελέγχου, της ελεγξιμότητας. Η διαφάνεια πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι εύληπτο, κατανοητό. Ποιο είναι το όφελος αν όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες, όμως ε, όταν αυτά όλα καταποντίζονται σε σχέση με τα ταμπού της πληροφορικής ή της πληροφόρησης. Θέτω ένα ερώτημα να μου αποσαφηνίσουν και μου στέλνουν 10 τόνους χαρτί με στοιχεία και με καταβυθίζουν. Και η προσέγγιση σε σχέση με τον όρο γραφειοκρατίας, γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Όλα αυτά η γραφειοκρατική επιβάρυνση ε, παρακολύουν το έργο μας και μας δυσχεραίνουν. Για παράδειγμα, να έχουμε ευληπτό χαρακτήρα σε σχέση με αυτές τις δράσεις. Θα συμφωνούσα αμέσως. Καλό θα ήταν να γνωρίζουμε σε σχέση με την ε, ανεξαρτησία ποιοι είναι οι ανεξάρτητοι. Δεν θα είχα καμιά αντίρρηση να καταχωρήσω τα ονόματα εκείνων με τους οποίους συνομιλώ. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε σε σχέση με την αξιολόγηση των ε, πληροφοριών η αξιολόγηση είναι σημαντικό ε, στοιχείο. Τα όρια, η αξιολόγηση, η αξιοποίηση είναι σημαντικά στοιχεία γοργότερα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Αν συμφωνούσαμε από αυτόν, γοργότερα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε σχέση με την επίτευξη των στόχων μας. Η σημαντική ανταλλαγή όμως των ε, στοιχείων να μην γίνεται εκτός δεδομένων πλαισίων γιατί δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας τότε. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές φορές ε, βρισκόμαστε σε αυτήν πολύ πιο μπρος από κράτη-μέλη και ίσως θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε πιο αποδοτικά. Σα ευχαριστώ πολύ και πολύ χρόνο αναλώνουμε και παρακαλώ λοιπόν να δοθούν οι απαντήσεις από τους πραγματογνώμονες. Είναι περιορισμένος ο χρόνος. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Έχετε εσείς πρώτος τον λόγο παρακαλώ. Ähm, Στον συνάδελφο μπορώ να προσθέσω κάποια στοιχεία λέει ο κύριος Βίλαντ. Αυτή τη μελέτη εδώ μόνο επιτροχά δεν μπόρεσα να την ε, διαβάσω αλλά μου λείπει, απουσιάζει πρέπει να πω εδώ, το ότι θα πρέπει επιστημονικά να δούμε ποια είναι τα επιχειρήματα του ότι κάποια θέματα πρέπει να έχουν, να εμπιστευτικό χαρακτήρα για κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι κυρία συνάδελφε Άουκεν, σας άκουσα πολύ νυφάλια και προσεκτικά. Ακούστε κι εσείς εμένα. Το σημείο είναι ότι γνωρίζω ιστορικούς που λένε ότι για δύο λόγους τα αρχεία των τελευταίων 30 ετών δεν είναι τόσο περιεκτικά όσο και παλαιότερα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα και διαγράφονται στη συνέχεια, εξαλείφονται και υπάρχουν άλλα θέματα στα οποία η καταγραφή τους, δηλαδή η, το ισχυρό σημείο της Ένωσης ήταν ότι μετά από 30-40 χρόνια μπορεί κανείς να δει για ποιον λόγο λήφθηκαν οι μένοι ή δε αποφάσεις. Να μην απουσιάσει αυτό το ισχυρό σημείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαλειφθεί. Έχω την εντύπωση ότι θα καταλήξουμε σε μια συλλογική άνοια ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι αρνητικό σημείο, είναι ευάλωτο σημείο, τροτό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> θα πρέπει σε σχέση με την καλύτερη διαφάνεια να υπάρχει απέναντί της η καλή διαχείριση, η χρηστή διαχείριση. Και θα έπρεπε έτσι λοιπόν οι ιστορικοί με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουν το θέμα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ρίγκαν παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Για την υποστήριξη των ε, Ευρωβουλευτών, όπως αναφέρθηκε, είναι πολύ σημαντικό για την αποτελεσματικότητα και του αξιώματος ε, του διαμεσολαβητού. Για τα θέματα αυτά πρέπει να θυμόμαστε το θέμα πρόσβασης σε έγγραφα θα είναι όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα στο μέλλον όταν οι χημικές δοκιμές και δοκιμασίες που θα γίνονται, που θα εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, θα αρχίσουν να ισχύουν. Όταν οι κλινικές δοκιμές σε σχέση με, αυτά, με αυτές τις ουσίες ε, θα ε, λειτουργούν και θα εφαρμόζονται έτσι και επειδή φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες του Ευρωκοινοβουλίου ότι συγκεκριμένοι κανόνες που αφορούν πρόσβαση σε παρόμοια τέτοια έγγραφα θα συμπεριλαμβάνουν υπό αυτό το πλαίσιο κανονισμού και κανόνες και διατάξεις που είναι πιο προοδευτικές και προοδευτικοί από ό,τι προβλέπεται στον κανονισμό 1049 Προφανώς υποστηρίζουμε την άποψη ότι αυτό είναι τεράστια σπουδαιότητα για τους πολίτες μας και αυτό αναφέρεται και στην απόφασή μας ο λίγων εβδομάδων ε, πριν. Θα είναι και πιο σημαντικό στο μέλλον όταν αυτά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων θα ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Δεύτερη παρατήρηση, εδώ δεν κάνουμε μόνο λόγο για πρόσβαση σε έγγραφα. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά θεμάτων σε πρόσβαση όσον αφορά τη διαφάνεια ομάδων πραγματογνωμόνων, ε, θέματα που αφορούν ε, αντικρώμενα συμφέροντα, ε, όλα αυτά συνδέονται με τα θέματα της διαφάνειας και από πλευράς διαμεσολαβητού συνεχίζεται το έργο σε αυτούς τους τομείς για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει εμπιστοσύνη στις δημόσιες αρχές και στον τρόπο λειτουργίας τους. Τελευταία παρατήρηση, σχεδιαζόμενη, σχεδιασμένη, προγραμματισμένη διαφάνεια. Γνωρίζουμε τις δυσχέρειες ε, όσον αφορά την ε, αντιμετώπιση πληροφοριών. Θα πρέπει οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαφάνεια εύληπτα και αποτελεσματικά. Είναι πολύ σημαντικό και οι αρχές να μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτό το μεγάλο όγκο ετοιμάτων και πληροφοριών με διαφάνεια, με σχεδιασμένο, προγραμματισμένο τρόπο για τράπεζες δεδομένων και διεργασίες, με τέτοιο τρόπο που εκ των υστέρων να μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα πρόσβασης για τους πολίτες η ε, αρχή και οι πολίτες να έχουν καλύτερη πρόσβαση ευχαριστώ. τελικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντάρμπισερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε... Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση της ε, Μαργκρέτε Άουκεν. Τι συγκεκριμένα μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Τρία πράγματα. Καταρχάς, ε, να συνεχίσει τη συνεργασία όπως γίνεται εδώ σήμερα με την κοινωνία των πολιτών, με τους πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες, ε, με το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας ε, για να προωθήσει την ε, διαφάνεια. Όσον αφορά το, τις ε, ταχυδρομικές διευθύνσεις, να απαντήσω στην Χάιντι Χάουτα, αλλά μας, μας ε, βοήθησαν διάφοροι για να καταλάβουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής, Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό. Όσον αφορά τους ε, πρόσφυγες, ε, πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσαν ότι γίνονταν κάποιες συζητήσεις σχετικά με την νομιμότητα ή όχι όσων συμβαίνουν. Το δεύτερο σημείο λοιπόν είναι ότι είναι σημαντικό να είναι κανείς υπόδειγμα διαφάνειας. Μπορώ να αναφέρω κάποιες περιπτώσεις όπου δεν ισχύει αυτό. Για παράδειγμα, όταν ζητήσαμε στοιχεία για τις δαπάνες της Κομισιόν ή ε, την προσφυγή στο δικαστήριο για τις δαπάνες των Ευρωβουλευτών. Ίσως θα μπορούσατε να το εξετάσετε αυτό. Και τέλος, ε, η τρίτη μου σύσταση είναι το Κοινοβούλιο να εξετάσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη όσον αφορά τη διαφάνεια, διότι ε, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις. Η Σουηδία και η Φιλανδία γιορτάζουν τώρα 250 χρόνια ε, καθεστώτος διαφάνειας, ενώ η Ιταλία έχει πολύ ε, ασθενές καθεστώς. Ε, ο, ο Ισπανικός νόμος δεν είναι πολύ καλός, ο, ο Ελληνικός είναι κακός. Ε. υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορές. Δεν είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους κανόνες διαφάνειας Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν αυξήσουμε ε, το επίπεδο και την κατανόηση στα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι μέρος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.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 to Ευχαριστώ. Θα ήθελα παρακαλώ να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι, γιατί δεν έχουμε πια χρόνο. Ευχαριστώ, πολύ σύντομα. Η Ολλανδική Προεδρία μίλησε για τις δυνατότητε ε, και το υπογραμμίζω αυτό, και έχει θετική στάση απέναντι στη διαφάνεια. Για τον 1049 υπάρχει μικρό περιθώριο να ξανανοίξουν οι διαπραγματεύσει. Ακόμα και η λισαβονοποίηση του κανονισμού, ε, που είναι κάτι που όλα τα θεσμικά όργανα θέλουν, δεν ήταν εφικτό να γίνει κάτι διάρκεια τη ε, Προεδρία μα. Για το Ευρωπαϊκό ε, Διοικητικό Δίκαιο, φυσικά το, εδώ το Συμβούλιο είναι στα χέρια τη Κομισιόν. Η Κομισιόν πρέπει πρώτα να κάνει μια πρόταση για να ξεκινήσουν οι συζητήσει στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους για την πρωινή ακρόασή μας, για τη συμμετοχή σας, για τις παρουσιάσεις σας, τις ομιλίες σας. Να κάνω μια σύντομη σύνοψη του τι ακούσαμε. Καταρχάς σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στην, ε, στα όσα κάνει η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η συνεισφορά του γραφείου του Διαμεσολαβητή στην, ε, στο χτίσιμο, στην οικοδόμηση αυτή της ε, διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεύτερον, πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι οι πολίτες αφυπνίζονται σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους για ενημέρωση. Αυτή η συνειδητοποίηση των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί εν συνεχεία από τη συνειδητοποίηση θα περάσουμε στην πίεση που θα ασκήσουν οι πολίτε στα δημόσια όργανα και στου δημόσιου φορεί για να λάβουν υπόψη τι ανάγκε τους. Μια καλή δημόσια ενημέρωση συνεισφέρει και στην αύξηση της ε, εμπιστοσύνη απέναντι στα θεσμικά όργανα. Μια σημαντική παρατήρηση ενό ε, Ευρωβουλευτή ήταν τα όρια αυτής της διαφάνεια. Υπάρχουν όρια στη διαφάνεια και αν ναι, πού θα πρέπει να θέσουμε αυτά τα όρια που παραδόξω θα πρέπει να τεθούν και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχουν διάφορα διλήμματα εδώ, διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και θα τα συζητήσουμε. Σίγουρα θα υπάρξουν ε, αντιμαχίες, θα υπάρξουν πολεμικές, ε, αντικρουόμενες απόψεις. Καταρχάς, ε, θα υπάρξουν συζητήσει για του ορισμού όλων αυτών των ενιών που συζήτησαμε σήμερα. Σα ευχαριστώ ακόμα μια φορά για αυτή τη συζήτηση και θα συνεχίσουμε σήμερα το απόγευμα.